Uh, Καλησπέρα σας ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε. Σημείο πρώτο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ως συνήθως ε, μεταδίδεται και από το διαδίκτυο απευθείας η συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να σας προτείνω δύο αλλαγές. Μετά το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, την γνωμοδότηση της κυρίας Σιλβί Γκουλάρ, ε, θα συζητήσουμε τα σημεία 9, 10 και 11. Και μετά το 11 θα επανέλθουμε στο 7 και 8. Αυτό ζήτησαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι οι εισηγητές. Άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι η συζήτησή μας για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα γίνει δημοσίω και όχι και κλεισμένο των θυρών όπως αρχικά προβλεπόταν. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Αν όχι να την εγκρίνουμε. Στο σημείο 2... Το δικό σας θέμα με τη και της Mercedes Μπρέσο μου ζήτησαν να το αλλάξουμε σειρά. Uh, Η γραμματεία έλαβε σχετικό αίτημα από την uh, κυρία Μπρέσο και είπε ότι τα είχατε συμφωνήσει, ότι είχατε συνεννοηθεί. Τι να κάνουμε, θα την ψάξουμε για να το διευκρινίσουμε. Μήπως είναι παρόν ε, κάποιος βοηθός της κυρίας Μπρέσο για να επικοινωνήσει μαζί της και να διαλευκάνουμε το θέμα. Θα το διευκρινίσουμε, Έλμαρ, για να δούμε αν υπάρχει λύση. Σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων ε, του Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Αν δεν υποβληθούν μέχρι το τέλος συνεδρίασης παρατηρήσεις θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Στο σημείο 4 στις δηλώσεις της Προέδρου, ανακοινώσει, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αποφασίστηκε από τους συντονιστές με κάποια καθυστέρηση οι για την μεταρρύθμιση του εκλογικού δικαίου να είναι η Ντανούτα Χίμπνερ και ο Γιώργο Λάινεν από το ΕΛΚ και του Σοσιαλιστές και Δημοκράτες αντίστοιχα. Επίσης σα εκπροσώπησα στην συνεδρίαση της ΚΟΖΑΚ, στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση της Ολομέλεια της ΚΟΖΑΚ που θα γίνει στη Ρήγα ε, το Μάιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ζήτησαν ε, μεγαλύτερη συμμετοχή στην ε, ευρωπαϊκή διαδικασία χάραξης πολιτικών. Θα συζητήσουμε και την συνεργασία μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπου θα γίνει και πιο διεξοδική ενημέρωση για τη θέση των Εθνικών Κοινοβουλίων και την προθυμία και την επιθυμία τους για στενότερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συμπράττουν πιο ενεργά στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα σημερινές αποφάσεις των συντονιστών. Οι συντονιστές ε, αποφάσισαν για τις ακροάσεις που αφορούν τα θεσμι... τις θεσμικές πτυχές των νέων κανόνων διακυβέρνησης να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Οικονομικών και να γίνει η ακρόαση στις 5 Μαΐου. Ελπίζω στις 11 Μαρτίου θα επικυρώσουν την ημερομηνία και οι συντονιστές της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Είναι η δεύτερη ημερομηνία που προτείνουμε. Επίσης, αν δεν βολεύει αυτή η ημερομηνία την Επιτροπή ΕΚΟΝ, θα την οργανώσουμε από μόνοι μας την δημόσια αυτή ακρόαση στις 5 Μαΐου. Άλλο θέμα που εξέτασαν οι συντονιστές είναι η πρόθεσή τους να οργανώσουν σεμινάριο για συγκριτικές ρυθμιστικές πρακτικές στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που ίσως ξεκινήσουν το καλοκαίρι για καλύτερη διοργανική συμφωνία για το εφνομοθετήν. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει το σεμινάριο τον Ιούνιο. Ζητήσαμε από το Τμήμα Πολιτικών να οργανώσει σχετικό σεμινάριο για τις ρυθμιστικές πρακτικές ή κανονιστικές πρακτικές. Επίσης προτάθηκε έκθεση πρωτοβουλίας από συνάδελφο της Γκουε που έγινε πια και υπουργό ε, στην Ελλάδα, τον κύριο Κατρούγκαλο. Ο κύριος Κατρούγκαλος είχε προτείνει έκθεση για τις θεσμικές πτυχές της οικονομικής διακυβέρνησης ως έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Αλλά δυστυχώς δεν τα βρήκαμε με την ΕΚΟΝ ε, ως προς τον τίτλο της έκθεσης στη διάσκεψη των ε, Προέδρων Επιτροπών Οπότε αποφασίσαμε να εστιάσουμε την έκθεση όχι σε εμφανή οικονομικά θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση. Βέβαια δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε πλήρως, αλλά λέμε για τη διεύρυνση οικονομικής, δημοκρατικής λογοδοσίας ε, και οικονομικές προκλήσεις ε, της διακυβέρνησης. και θα αντικατασταθεί ο κύριος Κατρούγκαλος από τον κύριο Χρυσόγωνο, αν ακούσαμε καλά την πρόεδρο. Επίσης, έμειναν και κάποιες εκκρεμότητες. Το αίτημα των Ιταλών, για παράδειγμα, για τη διευκρίνηση της νομικής κατάστασης σε σχέση με την νομοθεσία Σεβερίνο. Το συζητήσαμε με την νομική υπηρεσία και μας πρότεινε να περιμένουμε. Γιατί κρεμοδική παρόμοια υπόθεση στο, και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε περιμένουμε τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις και κατόπιν θα ενημερώσουμε τους Ιταλούς συναδέλφους. Επίσης, συμφωνήσαμε να γνωμοδοτήσουμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το περίφημο επενδυτικό σχέδιο του κυρίου Γιούγκερ. Τη σχετική γνωμοδότηση την ανέλαβε μέλος του ΕΛΚ. Αυτά ως προς το 5 της ανακοινώσεις της Προέδρου και περνάμε στο 6 τη γνωμοδότηση της ε, Σιλβί Γκουλάρ. Έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και τώρα έχει και πάλι το λόγο Σιλβί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τους ε, Shadow και όλους αυτούς που συνεισέφεραν με τροπολογίες επί τη διαδικασίας, επί τη μεθόδου μάλλον. Στην έκθεση ΑΦΚΟ είμαστε πιο δυνατοί όσο επικεντρωνόμαστε στα συνταγματικά θέματα, στα θέματα δικαίου. Και υπό το πνεύμα αυτό θα σας πρότεινα αυτές τις συμβαστικές ε, τροπολογίες και θα ήθελα να σημειώσω για αυτούς που δεν ήταν εκεί ότι ο κύριος Ντράγκη είπε στην Ολομέλεια ότι θα επανεκκινήσει η άσκηση των τεσσάρων προέδρων που είχε καταλήξει σε μια πρώτη έκθεση σχετικά με τον κύριο Φαν ε, και είχε ζητήσει από το κοινοβούλιο ο κύριος Ντράγκη να συνεισφέρει σε μια βελτίωση, σε μια βελτιωτική προσπάθεια για να φτάσουμε σε μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Τώρα σύντομα επειδή δεν έχουμε χρόνο και ελπίζω πρόεδρε οι Σάντο να παρέμβουν γιατί την περασμένη φορά δεν είχαμε χρόνο έχουμε κάποια σημεία συγκλήσεως και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σχετικά με την αύξηση της ε, ευθύνης της λογοδοσίας σχετικά με τις αποφάσεις έχουμε κάποιες ενισχύσεις της ε, ενωσιακής μεθόδου ε, για τα διακυβερνητικά και την εσωμάτωσή τους στην ε, συνθήκη για την αύξηση και την ενίσχυση της δημοκρατίας σε σχέση με το γεγονό ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ενέχονται πολύ περισσότερο σε κάποιες διαδικασίες που άπτουν τις θερμοδιότητες τους ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγγυάται την ε, λογοδοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκεί έχουμε σύγκληση, διομαδικά, πολιτικά. Πρέπει να δούμε για τις επενδύσεις, στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις ε, ε, δαπάνες και θεωρώ πολύ πιο επικοδομητικό να, δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ακολουθούμε τους κανόνες παρά να φανταζόμαστε θεωρητικές ευελιξίες που τελικά σημαίνουν παράκαμψη των κανόνων. Επίσης υπάρχει ένα θέμα που νομίζω ότι τίθεται αρκετά συχνά στην Επιτροπή, για παράδειγμα την έκθεση του κυρίου Γουαλτιέρη για την ε, multi-tier governance, πρέπει να μιλήσουμε για τροποποίηση των συνδικών ή όχι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ναι, αλλά Βεβαίω πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα περιθώρια που, είναι, που έχουμε στη θέση μας. Δεν πρέπει να φοβηθούμε ε, κάποιους ε, προσανατολισμούς. Έχουμε και ένα σημείωμα αναλυτικό του κυρίου Γιούνκερ ε, από, τι τις 12 Φεβρουαρίου, υπάρχει μια σημείωση του κυρίου Ντράγκη, υπάρχει μια δουλειά στην οποία εγγράφεται το Κοινοβούλιο, ο κύριος Σούλτς έχει πει ότι θα διαματήσει ένα ρόλο, αλλά η εντολή Εντό τη οποία θα πρέπει να εμπνεύσει τη δουλειά των τεσσάρων προάδρων ε, το κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι μέσω των επιτροπών. Άρα ας μην διστάσουμε να το εξετάσουμε αυτό το θέμα σε ό,τι με αφορά και ελπίζω εδώ να σας πείσω λίγο λίγο για την ένωση την οικονομική και την νομισματική ε, σε ό,τι αφορά παρεκκλήσεις ε, από το υπόλοιπο ενωσιακό δίκαιο και είναι η συνθήκη που το λέω και εγώ δεν είναι σε ένα κράτος δικαίου που θέλουμε να υπάρχουν κοινών, ε, κανόνες τις οποίες θα τους σεβόμαστε. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να αγνοούμε απολύτως το, το δικαστήριο και για να μην έχουμε παρανοήσεις. Ε, στην συνθήκη έχουμε, έχουμε προσφυγές σε παραλήψη αλλά έχουμε και προσφυγές για προσακύρωση. Δηλαδή, σήμερα το βλέπουμε με την αύξηση της ισχύω της Τρόικα, για παράδειγμα, η οποία δεν είχε νομική βάση αγκύρωση στη συνθήκη, γιατί τότε αν είχε θα μπορούσε κανείς να είχε εκφράσει μια διαφωνία. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ένα κράτος δικαίου λοιπόν δεν πρέπει να φοβάται να χρησιμοποιήσει όλες τις διόδους προσφυγής, το οποίο δεν σημαίνει και επαναλαμβάνω, ότι θα αντικαταστήσουμε τη δικαστική εξουσία από την πολιτική ηγεσία. Υπό, την, υπό τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας έχουμε συντάγματα, έχουμε χώρες όπως η Γερμανία αλλά και άλλες όπου το συνταγματικό δικαστήριο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Επομένως, στην Επιτροπή μας με όλες τις επιφυλάξεις για το μέσο και μάκρο πρόθεσμο πλαίσιο, πρέπει να θίξουμε το θέμα αυτού του μη πλήρους κράτους δικαίου. Και αυτή η συζήτηση επί της Ένωσης ε, της Οικονομικής και της ε, Νομισματικής ε, κυνηγάει την ουρά της εδώ και πολλά χρόνια και πρέπει να, να αποφύγουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια προκειμένου να πείσουμε κάποιον στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε την ευρέα τη δυνατή ε, συνένεση και πλειοψηφία Αυτά είχα να σα πω. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σιλβί, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ο Έλμαρ Μπρόκ ε, για το ΕΛΚ, ε, νομίζω. Για τους Σάντου ε, θέλετε κι εσείς να πείτε κάτι ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σιλβί Γκουλάρ για την έκθεση αυτή. Νομίζω πως είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαρίσει και να δει η Επιτροπή. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Βεβαίως ε, της δικός μας Επιτροπής το έργο είναι να δούμε το θεσμικό πλαίσιο, τι γίνεται και πιθανώς αν χρειάζονται κάποιες αλλαγές στην ε, συνθήκη. Και δεν είναι θέμα τόσο ζήτημα της κοινωνικο-οικονομικής, ε, του κοινωνικο-οικονομικού προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι αυτή η δικιά μας η δουλειά. Αυτό το έχουμε συζητήσει και στην έκθεση Μπρέσο Μπροκ Φερχόφστατ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα εμείς τη συζήτηση αν πρέπει να πάμε περισσότερο προς την πτυχή την κοινωνική, της ανταγωνιστικότητας, δεν είναι αυτή η δικιά μας η δουλειά εδώ πέρα. Πρέπει να διαπιστώσουμε όμως με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ξεπεράσουμε την κρίση και πώς θα μπορέσουν να ενταχθούν στο κοινοτικό δίκαιο και να μην είναι διακυβερνητικά εντελώ, τα ζητήματα που έχουν να κάνει με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και βεβαίω. ξεκαθαρίζουμε με ποιον τρόπο παραμερίζονται τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην διαδικασία αυτή. Αυτά μου φαίνονται εμένα ότι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Τώρα η ουσία αναφέρεται στην συνθήκη. Έχουμε άρθρο που αφορά και την ανταγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη και την ε, κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά αυτά δεν έχουν ε, τόση σημασία εδώ πέρα. Νομίζω πως υπάρχει ούτως ή άλλως πάντως μια σαφής αφετηρία στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας η οποία είναι τελείως ισορροπημένη και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή. Νομίζω πως αυτό είναι σαφές. Για μένα είναι σημαντικό αυτό το θέμα, πιο δηλαδή, ότι πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την ισορροπία μεταξύ ε, υγιών οικονομικών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης. Αν μπορέσουμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό και να αποδείξουμε πώς οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βοηθούν την ανάπτυξη και πώς θα μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Να πω επίσης πως ε, έχω καταθέσει μια τροπολογία που συμπληρώνει αυτά τα οποία λέει η κυρία Γκουλάρα σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τα είχαμε πει αυτά και στο έγγραφο του Φανδόμποη. Ότι δηλαδή όταν καταρτίζονται οι ετήσιες συστάσει αναχώρα στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης ανάπτυξη δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις κατευθυντήριες γραμμές. Και θεωρώ πως η Κομισιόν θα πρέπει να δεσμεύεται οι κατευθυντήριε αυτές γραμμές να είναι αποτέλεσμα συναπόφασης και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ισχύουν 4-5 χρόνια ε, στις οποίες θα αναφέρονται αρχές και θα καθορίζεται ξεκάθαρα ε, ποιοι τομείς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η αδυναμία αυτών των στάσεων είναι πως ασχολούνται με χίλια θέματα που κανέναν δεν ενδιαφέρουν και άρα δεν έχει την απαραίτητη όθηση για να προωθήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει λοιπόν να επικεντρώνονται σε πέντε σημαντικά πράγματα. Αυτό μπορεί να γίνει επί στην έκονα, αλλά μπορούμε νομίζω και εμείς να το πούμε. Αλλά θεωρώ πως οι κατευθυντήρες γραμμές πρέπει να είναι αποτέλεσμα συναπόφασης. Και εάν με βάση αυτές τις συστάσεις βγάλουν μετά τα συμπεράσματά τους ε, τα κράτη Δηλαδή, με ποιον τρόπο σκέφτονται να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα που προτείνονται στις συστάσεις, τότε θεωρούμε πως πρέπει να λυθούν υπόψη δύο πράγματα. Πρώτον, σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει κίνητρα χωρίς να οδηγηθούμε σε έναν λεγόμενο ηθικό κίνδυνο, ε, αλλά κάποια κίνητρα είτε μέσω των περιφερειακών κονδυλίων ε, για να υπάρξει μία βοήθεια από πλευράς Ευρώπης για την ε, αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας για να υπάρξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στο μης στους οποίους υπάρχουν εθνικές αρμοδιότητες. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις τα θέματα αυτά τα οποία αναφέρονται είναι εθνική αρμοδιότητα. Αγορά εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, ζητήματα απεργιών. Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή αρμοδιότητα σε αυτά τα θέματα. Αλλά με ποιο τρόπο μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κίνητρα για αυτά τα ζητήματα. Και επειδή είναι όντω εθνικές υποθέσεις πρέπει να συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Όταν προτείνει μια χώρα λοιπόν ένα εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να έχει βεβαίως και τη στήριξη του ε, Εθνικού Κοινοβουλίου. Και έτσι θα έχουμε κοινοβουλευτική συμμετοχή και στα δύο επίπεδα. Και νομίζω έτσι ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα οποία λέει η κυρία Γκουλάρ. Να μην έχουμε δηλαδή μικτές αρμοδιότητες, αλλά ο καθένας να είναι υπεύθυνος στο επίπεδό του. Εμένα δεν αρέσει καθόλου αυτό το, αυτή η κοινή ε, συνέλευση που γίνεται με βάση το άρθρο 13. Δεν αλλάζουν οι αρμοδιότητες. Σε ένα επίπεδο λαμβάνεται η απόφαση και αυτή πρέπει να είναι υπεύθυνη οι συστάσεις γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα πρέπει να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εφαρμογή του προγράμματος είναι εθνική νομοθεσία, οπότε εκεί πέρα πρέπει να μπουν τα εθνικά κοινοβούλια. Με μια τέτοια δομή νομίζω θα αποφύγουμε βεβαίως και την δυσπιστία από πλευράς εθνικών κοινοβουλίων. και έτσι νομίζω πως ε, θα έχουμε και ένα υψηλότερο βαθμό νομιμοποίησης. Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς όπως είπα να ενισχυθεί αυτή η νομοποίηση. Επίσης να πω πως δυστυχώς ε, κατέθεσα και κατά λάθο μια τροπολογία την οποία αποσύρω αυτή που λέει να διαγραφεί το άρθρο για τη συμμετοχή του δικαστηρίου. Ε, πρόκειται για... Για έγινε μια ανάλογη προσπάθεια και στην ε, συνέλευση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα χώρο χωρίς ε, δίκαιο και τότε απέτυχε και τώρα βεβαίως το ζήτημα δεν μπορεί να μην είναι αρμόδιο το 10 και νομίζω πως αυτά που λέω θα ικανοποιήσουν και την κυρία Γκουλάρα και μπορούμε να συνοηθούμε νομίζω με την σοσιαλδημοκρατική ομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θεωρώ σωστά αλλά όπως είπα κάποια άλλα είναι τελείως οικονομικά και όχι τόσο συνταγματικά. Μια άλλη ιδέα που είναι ενδιαφέρουσα ε, την οποία ανέφερε η κυρία Γκουλάρ έχει σχέση με τον ορισμό των επενδυτικών δαπανών και των λοιπόν δαπανών. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να δούμε το όριο του χρέους όπως αυτό είναι στο Μαστίχ και να γίνει μια διάκριση μεταξύ των ε, δαπανών. Τα χρέη όμως είναι χρέη, ε, ανεξαρτήτως του τι τα κάνουμε τα λεφτά. Και αν ε, καταλήξουμε σε μια θέση ότι δεν ισχύει ο κανόνας επειδή κάποιες δαπάνες είναι επενδύσεις, τι θα γίνει, θα έχουμε πάλι δαπάνες καταναλωτικές οι οποίες θα δηλώνονται ως ε, επενδυτικές. Αλλά Γενικότερα όμω για λόγους αξιοπιστίας ενός προϋπολογισμού ανεξαρτήτως από το όριο του χρέους πράγματι πρέπει να δούμε το ποσοστό επενδυτικών και μη δαπανών γιατί βεβαίως ένας προπολογισμό με περισσότερες επενδυτικές δαπάνες είναι πιο ε, θετικός ε, και για το μέλλον. Και μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους των σοσιαλιστών ο κύριος Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν ε, να ευχαριστήσω θερμά την εισηγητριά μας, την κυρία Σιλβί Γκουλάρ, για την προθυμία της ε, να αναζητήσει συμβαστικές ε, λύσεις για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και να εξασφαλίσει συνεννόηση μεταξύ των σχεδόν εισηγητών. Θα ήθελα να τη διαβεβαιώσω ότι η σοσιαλιστική ομάδα είναι πρόθυμη να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια ανέβρεσης συμβαστικών προτάσεων και λύσεων. Θα ήθελα επ' να πω ότι συμφωνώ με τις βασικές παρατηρήσεις της συγκεντρίας. Δηλαδή αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Δηλαδή κυρίως σε θεσμικά και συνταγματικά θέματα θα πρέπει να επικεντρωθεί η Επιτροπή μας. Επίσης θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή, Εκών, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια κατ' ουσία και στην ε, εισηγήτρια αυτής της Επιτροπής, της ΕΚΟΝ, την κυρία Περβάνς Περές, Μπερές που έχει αναλάβει την εκπόνηση της κυρίας έκθεσης. Εμείς ε, Καταθέσαμε πολλές τροπολογίες. Μπορώ να σας πω ότι εμείς καταθέσαμε όλες σχεδόν τις τροπολογίες από τις 42 που κατατέθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε αρνητικοί απέναντι στην ε, ανέβρεση συμβαστικών λύσεων. Εμείς θέλουμε κυρίως να επισημάνουμε τα ουσιώδη στοιχεία αυτού του σχεδίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και να επισημάνουμε το γεγονός ότι η ΟΝΕ στερείται μηχανισμών που να εξασφαλίζουν ε, δημοσιονομική ικανότητα, τεχνική, ε, χρηματοοικονομική αρρωγή και ένα, στερείται και ενός θεσμικού πυλώνα και άρα πυλώνα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Δυστυχώς εκεί χωλαίνει η όλη διαδικασία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η έλλειψη, στην έλλειψη της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Γι' αυτό και συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ΟΝΕ, όπως προτείνει και η συγγήτρια. Και το μεγαλύτερο τμήμα των προτάσεών μας αυτό το στόχο έχει. Δηλαδή, θέλουμε να διευκρινίσουμε την ενισχυμένη συμβολή που περιμέναμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εγγυηθούμε ακριβώς τη δημοκρατική νομοποίηση της οικονομικής διακυβέρνησης. Μία άλλη ανησυχία μας αφορά τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται οι κανόνες στο κοινοτικό, ε, στην κοινοτική ένωμη τάξη στο κοινοτικό νομικό σύστημα. Όπως είπε η κυρία Κουλάρ, θα πρέπει να βρούμε τρόπους και μηχανισμούς για να αναβαθμίσουμε την κοινοτική μέθοδο και επίσης να είμαστε πιο φιλόδοξοι στον τρόπο ερμηνείας της δημοσιονομικής ελαστικότητας ή της δημοσιονομικής ευελιξίας. Αν δεν κάνω λάθος, ε, εντός ολίγου θα συνεδριάσουν οι σκιώδεις συγητές μαζί με την εισηγήτρια. Εκεί θα παρουσιάσω τις τροπολογίες μου και σας διαβεβαιώ ότι είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε συμβαστικές λύσεις. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που επισημάνατε πριν από λίγο είναι να δούμε αν χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία, περισσότερη ελευθερία, χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο τάσεων. Γιατί συνήθως οι κανόνες και κυρίως οι κανόνες της δημοσιονομικής πολιτικής και της ε, οικονομικής διακυβέρνησης αφήνουν ένα περιθώριο ελιγμών, αφήνουν μια ελαστικότητα στη δημοσιονομική πολιτική. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να αξιοποιήσουμε τους υπάρχοντες κανόνες να και να αξιοποιήσουμε την ευελιξία πολύ περισσότερο από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα γιατί η δυνατότητα υπάρχει. Και ουσιαστικά αυτό αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της και κάνει και κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι η ευελιξία αντιστρατεύεται τους κανόνες. Αντίθετα θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό ευελιξίας που εμπεριέχεται στους δημοσιονομικούς κανόνες. Επίσης, Υπάρχουν και κάποιες νομικές εδώ παρατηρήσεις. Η δημοσιονομική ευελιξία, κυρίως ό,τι αφορά την εφαρμογή της ρήτρα των επενδύσεων, θα πρέπει να επανεξεταστεί, να αναθεωρηθεί, ώστε να ισχύει και για αυτό το διορθωτικό ε, μηχανισμό ή το διορθωτικό βραχίωνα του συμφώνου. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα της αρχής της ισότητας. Είναι προφανές ότι οι χώρες που βρίσκονται στο προληπτικό βραχίωνα και εκείνες που βρίσκονται στον διορθωτικό βραχίωνα αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Και η επιτρεπόμενη διαφορετική μεταχείριση θα πρέπει να είναι ανάλογη με τις διαφορές Τίποτα δεν δικαιολογεί η συνεισφορά μιας χώρας στο ευρωπαϊκό σχέδιο. να αντιμετωπίζεται ως ε, ότι βρίσκεται στο απειρόβλητο της, ε, του συμφώνου. και αλλιώς να αντιμετωπίζεται η συμμετοχή στα κοινοτικά ταμεία και αλλιώς στην, στο κοινοτικό προϋπολογισμό. Γιατί έχουμε δύο διαφορετικούς ε, τρόπους επενδύσεων που παρόλο που αφορούν και οι δύο τις ε, κοινοτικές επενδύσεις αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Τέτοια διαφοροποιημένη μεταχείριση δεν δικαιολογείται κατά τη γνώμη μου σε τέτοιο βαθμό. Ιδιαίτερα μεταξύ του βραχίωρα, του προληπτικού και του διορθωτικού. Επειδή η ισότητα μα είναι ιδιαίτερη προσφυλή, θα θέλαμε να ισχύει πολύ περισσότερο και κατά την εφαρμογή της ελαστικότητας στη ρήτρα των επενδύσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των συνθήκων. Η Σιλβί Γκουλάρ προτείνει αναθεώρηση των συνθήκων και λέει ότι η δική μας επιτροπή, η συνταγματική επιτροπή είναι αρμόδια να συζητήσει την πιθανότητα αυτή. Αναφίβολα ένα τέτοιο θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Η πρόταση όμως που γίνεται αφορά μια χειρουργική αναθεώρηση και αφορά την ε, ανάμιξη των δικαστηρίων στην ε, εφαρμογή ε, ε, κυρώσεων, στην επιβολή κυρώσεων κατά τον παραβοτό, εφόσον γίνει προηγουμένω μια διάγνωση της παραβίασης των ε, δημοσιονομικών κανόνων. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, δεν συμμερίζεται αυτή την πρόταση. Γι' αυτό και θα προτείνουμε διαγραφή της παραγράφου 6. Ακόμη και με τη νέα διατύπωση που προτείνει η συγκήτρια το πρόβλημα δεν επιλύεται. Και αν θέλουμε να εξετάσουμε την αναθεώρηση των συνθήκων και μια αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης για να βελτιωθεί η δημοκρατική νομοποίηση, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι σε μια τέτοια συζήτηση. Και πιστεύω ότι με μια τέτοια ευρύτερη αναθεώρηση θα φέρναμε και καλύτερα αποτελέσματα στην οικονομική διακυβέρνηση. Παρακαλώ, αν μακρηγορείτε όλοι τόσο, δεν πρόκειται να καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε την ημερήσια διάταξη. Θα χρειαστεί να προτείνω να αφαιρεθούν κάποια σημεία από την ημερήσια διάταξη. Λυπάμαι που σας πιέζω, αλλά παρακαλώ να το λάβετε υπόψη. Ο κύριος Λούκα. No. Uh, Η κυρία Σπινέλη για τον ΚΟΕ. Όσο πιο σύντομα μπορείτε, παρακαλώ. Ναι, πρόεδρε. Ναι, ευχαριστήσω την κυρία Γκουλά και συμφωνώ μαζί της ότι δεν πρέπει να γυρίζουμε γύρω-γύρω από το θέμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την κοινωνική διάσταση της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι θεσμικό το θέμα της κοινωνικής διάτασης. Το λέω γιατί μιλούμε για τους προσανατολισμούς της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής και αν προσθέσει κανείς το επίθετο κοινωνική γίνεται αμέσως αυτόματα θεσμικά σχετικό. Η προσχώρηση λοιπόν στη χάρτα την ε, κοινωνική και η ιδέα που θα μπορούσε να έχει κανείς σχετικά με με ένα κοινωνικό μαζί με το Οικονομικό Συμβούλιο όπως ε, συμβαίνει στα λεγόμενα συμβούλια τζάμπο. Τώρα για την ακύρωση Τη Τρόικα ε, δεν έχω να προσθέσω και πολλά, ήδη το είπε το Κοινοβούλιο αυτό και να εκφράσω και κάποιες αμφιβολίες για την συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και του Πρόεδρου στην εργασία των τεσσάρων Πρόεδρων. Όχι υπό την έννοια ότι δεν θέλω να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο, αλλά προκειμένου το Κοινοβούλιο να είναι συνομιλητής και να μην έχει τα χέρια δεμένα ο κύριος Σούλτς από τους άλλους πρόεδρους. Αυτό. Μάλιστα Μπάρμπαρα, ευχαριστούμε. Ο, ο κύριος Ντιουγό είναι εδώ. Σύντομα αν θέλετε. Βεβαίως πρόεδρε θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Να πω, καταρχάς να Ευχαριστήσω τη Σιλβή για τη δουλειά και για την επιχειρηματολογία της και για το διάλογο που εγκαταστάθηκε. Τώρα, εγώ δυσκολεύομαι, εξακολουθώ να δυσκολεύομαι, ιδιαίτερα στο θεσμικό πλαίσιο να διακρίνω το οικονομικό από το κοινωνικό. Και θα έλεγα συνολικά ένα κοινοβούλιο δεν μπορεί να απομονώνει ορισμένα θέματα και να λέει αυτά είναι τεχνικά και τα άλλα είναι διανοητικά ή πνευματικά ή οτιδήποτε άλλο, όπως θέλουμε να το πούμε. Εγώ δεν εξελέγει από τους πολίτες ώστε να εφαρμόζω πιστά και τεχνικά κάποιες διατάξεις ή κανόνες και το λέω αυτό στη Σιλβή με όλο το σεβασμό και τη συμπάθεια που τις έχω. Αλλά σκέπτομαι ε, το εξής που θα ήθελα να υπογραμμίσω γιατί στα υπόλοιπα είμαι βέβαιος ότι συμφωνούμε. Το ε, θέμα του δικαστηρίου, το θέμα των κυρώσεων μη πολιτικής φύσεως, νομικής φύσεως των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες γιατί αυτό είναι το σημείο κίνησης τη όλη διαδικασία, του κύκλου των κυρώσεων, είναι ότι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Όλα αυτά θέτουν τα πάντα ένα αμφιβόλο. Εάν οι δημοσιονομικές πιέσεις έχουν γίνει αποδεκτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι γιατί ακριβώς ο έλεγχο ήταν πολιτικός ο Ασκήτο. Και λέμε, ναι, θα βάλουμε περιορισμούς δημοσιονομικούς, αλλά αυτούς τους περιορισμούς θα τους ξαναδούμε. Δηλαδή, τους αποδεχθήκατε, αλλά θα, και παράλληλα θα είμαστε και σε θέση να σας επιβάλλουμε κυρώσεις αν δεν ε, τηρείτε τους κανόνες. Δηλαδή, ε, θα έλεγα ότι είναι ζωτική σημασία το θέμα αυτό για την ανακοίνωση. Αν αυτό το δούμε καθαρά οικονομοτεχνικά, νομοτεχνικά, θα χάσουμε, θα απολέσουμε τη δυνατότητα εξέβρεση ισορροπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επ' αυτού συμφωνούμε απολύτως πιστεύω. Πρέπει να ξαναδώσουμε στο Κοινοβούλιο και γι' αυτό και εγώ δεν φοβάμαι καθόλου την θεσμική μεταρρύθμιση και, τη, και την, ε, και την επανεξέταση της συνθήκης. Πρέπει και το Eurogroup να μην μπορούν να θέτουν μόνοι τους τα όρια της ισχύω τους. Ε, να πω και εγώ ευχαριστώ σε όλους. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε μόνο το εξής, μία κουβέντα επί της ουσίας. Πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά δεν θέλω να καθυστερήσω τα πράγματα. Καταρχάς, δεν πρότεινα αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων νομοθετικών ή νομικών αναφέρθηκα στον κράτο δικαίου στην Ένωση, την Οικονομική και Νομισματική. Δεν μπορεί οι πολιτικές να είναι εκτός ενός θεσμικού πλαισίου, συνταγματικού πλαισίου, πλαισίου συνθήκων δηλαδή. Ο Πασκάλ έχει δίκιο. Υπάρχουν θέματα οικονομικά και κοινωνικά, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που υποσκάπτει τα πράγματα. Οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν δεσμεύσει και μετά δεν τι τηρούν. Επομένω, όπω και να το δει κανεί, είτε να πάμε υπερβολικά στο θέμα των κυρώσεων και το τεχνικό θέμα της, της Τρόικα, είτε το να το δούμε υπερβολικά ελαφρά την καρδία, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο, δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειε, αυτό ήθελα να διαφημίσω. Ναι, πρέπει να ψηφίσουμε 17 Μαρτίου. Επομένως, ε, λέει η Πρόεδρος, ελπίζω ότι Ακόμα και χωρίς τον έλεγχο του δικαστηρίου, Πρόεδρε, θα το κάνουμε, θα τα καταφέρουμε. Ωραία, πάμε στο σημείο 9. Γκονσάλες Πόνς ε, και η γνωμοδότηση για τη Συμφωνία Διατλαντικού Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, γνωρίζετε όλοι, εδώ και πολλές εβδομάδες ασχολούμαι με το σχέδιο έκθεσης, ε, με προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου που είναι αρμόδια επί τη ουσία ε, για την Συμφωνία TTIP, τη και Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων. Μετά από συναντήσεις που είχα και συνομιλήσει με τους σκιώδεις ηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων, κατέληξε σε ένα κείμενο που ευελπιστώ ότι θα βρει σύμφωνο στους συναδέλφους και περιλαμβάνει τις βασικές προτάσεις της Επιτροπή μας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Επειδή είμαστε ε, δεσμευμένοι από τον τύπο για τις γνωμοδότησεις αυτές, ε, περιλαμβάνουμε κάποιες αιτιολογικές σκέψεις που αναφέρονται στις αλλαγές που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνας ε, σε θέματα εξωτερικού εμπορίου. Γιατί χάρη στη συνθήκη αυτή επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής της κοινή εμπορικής πολιτικής ώστε να περιλαμβάνει και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Και έτσι το Κοινοβούλιο έχει νέε εξουσίες σε τέτοιου είδου συμφωνίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιμέρου σημεία της γνωμοδότηση, που την έχω ήδη υποβάλει και την έχετε λάβει όλοι οι συνάδελφοι, αναφέρεται ότι ακόμη και αν σε τέτοιου είδου διαπραγματεύσεις απαιτείται ένα βαθμό εμπιστευτικότητα για να είναι αποτελεσματικέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πρωτοπόρα σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση τη διαφάνεια. Γι' αυτό και εκτιμούμε την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει τις διαπραγματεύσεις πιο διαφανείς και προσιτές στο κοινό. Αναφέρονται και οι συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή της 6 Ιανουαρίου 2015 για να ενισχυθεί περαιτέρω η νομιμότητα και η διαφάνεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Αναφέρονται επίση ότι και τα, Ευρωπαϊκά κοινοβούλια, και τα Εθνικά Συγνώμη Κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν στη συμφωνία για το TTIP και να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να κληθούν ε, τα, τα Εθνικά Κοινοβούλια να κυρώσουν ε, την ε, συμφωνία αυτή αν θεωρηθεί ως συμφωνία μεικτού τύπου με ισχυρό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Πιστεύω ότι αν διεκπαιρεωθεί το TTIP θα είναι συμφωνία μεικτού τύπου. Οπότε πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει και τα εθνικά κοινοβούλια να αποφανθούν επί της συμφωνίας αυτής. Γι' αυτό και θα πρέπει να τα εμπλέξουμε σε πρόορη φάση της διαδικασίας και των διαπραγματεύσεων, ώστε να μην καταρρεύσει μια επιτυχής διαπραγμάτευση επειδή ένα εθνικό κοινοβούλιο αισθανθεί προσβεβλημένο από την περιθωριοποίηση και καταψηφίσει τη συμφωνία. Επίσης, ε, χαιρετίζει την ε, πρόταση Μητρώου Διαφάνειας ε, για τα λόμπι που παρίσταται στις διαπραγματεύσεις του TTIP, γιατί όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι ομάδες συμφερόντων οικονομικών και πολιτικών που εμπλέκονται στη διαδικασία και συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις TTIP. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες και τους κανονισμούς απέθυνα έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει το ρόλο που θα έχει το, το ρόλο και τη νομική υπόσταση που θα έχουν τα πορίσματα του λεγόμενου Ρυθμιστικού Συμβουλίου Συνεργασίας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το χαρακτήρα και τη νομική υπόσταση αυτών των πορισμάτων του Ρυθμιστικού Συμβουλίου Συνεργασίας και αν θα έχουν ή όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. Γιατί αν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, ε, τότε θα παραβιάζουν ε, την ε, νομοθεσία και τις ε, συνθήκες. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον γνωστό μηχανισμό ISDS, το Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή Κράτους. Θεωρούμε ότι ο μηχανισμός αυτός είναι κατάλληλο εργαλείο για την προστασία των επενδυτών και περιλαμβάνεται σε πολλές διεθνείς συμφωνίες. Θα πρέπει να προβλέπεται δίκαιη και μη διακριτική μεταχείριση των επενδύσεων. Αλλά θα ήθελα να δηλώσω ρητά και κατηγορηματικά ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να μην οριοθετεί, να μην περιορίζει, να μην υποσκάφτει τις δυνατότητες των εθνικών και τοπικών αρχών να νομοθετούν τις δικές τους πολιτικές, ιδιαίτερα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Και σε καμία περίπτωση ένας τέτοιος μηχανισμός επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους δεν μπορεί να αντίκειται ε, στο συνταγματικό δίκαιο ή να παραβιάζει ε, τη συνταγματικότητα και τη συνταγματική αναμετάξη των κρατών μέλων. Αυτές είναι οι προτάσεις της γνωμοδότησής μου. Περιμένω τις παρατηρήσεις ε, των σκιωδών εισηγητών και των πολιτικών ομάδων με πολύ προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πέντρο Σίλβα Περέρα, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή μας, τον κύριο Κωνσάλες Πόνς, ήδη έκανε πολλές προσπάθειες ε, συνενόησης με τις πολιτικές ομάδες για να καταλήξουμε σε ένα συνενετικό κείμενο. Ήδη συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να περάσουμε στην εξέταση των τροπολογιών και στην ανέβρεση συνένεσης ε, επί της γνωμοδοτήσεως. Εμείς συμφωνούμε με το ύφος και τον τόνο αυτής της γνωμοδότησης Αντιλαμβανόμαστε ε, τη μία του ISDS, του Μηχανισμού Επίλυσης Διαφορών Επένδυτη Κράτους. Ε, ε, θα θέλαμε μια αλλαγή της διατύπωσης της παραγράφου, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η συμπερίληψη αυτού του μηχανισμού επίλυσης των διαφορών στην, στις διαπραγματεύσεις και φυσικά συμφωνούμε με την έγκαιρη ανάμειξη των Εθνικών Κοινοβουλίων στις διαπραγματεύσεις και στην διαδικασία αυτή. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αρχή της συνοχής των πολιτικών. Επ' αυτού θα καταθέσουμε και τροπολογία. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες ε, για τον τρόπο που προτείνεται η σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας στο λόμπι. Δεν είμαστε κατά της αρχής, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να έχουμε ειδικό κανόνα ε, Μητρώου σε μια συγκεκριμένη διαπραγματευτική διαδικασία. Ως προς αυτό έχουμε κάποιες ανησυχίες. Πάντως με πολύ επικοδομητικό πνεύμα θα καταθέσουμε τις, προσπα... τις προτάσεις μας και τις τροπολογίες εν ώψη της ανέβρεσης ε, συνενετικής λύσης. Δεν ξέρω αν ο Μάρκος Κρέλτσερ είναι παρόν, όχι, ούτε ο Σαλ ούτε ο Σόλτς. Ο Πασκάλ Ντουιραν είναι εδώ. Ευχαριστώ. Ε, έχω την αίσθηση ότι μου δίνεται το λόγο από τους πρώτους. Δεν έχω συνηθίσει. Νομίζω ότι ήταν πολύ αντικειμενικό το έργο του συντάκτη της γνωμοδότησης και βάζει την Επιτροπή μας ε, σε ένα πολύ επικοδομητικό κλίμα για την σύνταξη της γνωμοδότησης και χωρίς να τροφοδοτεί καθόλου αντιπαραθέσεις και αψημαχίες. Λυπούμε που έχουμε διαφωνία ως, προ ISDS, ως προς το ISDS, το Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή κράτου. γιατί για τα κανονιστικά θέματα συμφωνούμε, στο θέμα της διαφάνειας και του Μητρώου επίσης συμφωνούμε, θεωρούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Το μόνο στοιχείο που μας ε, χωρίζει και θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει να το συζητήσουμε θα έχει ε, κεντρικό χαρακτήρα ε, στο κατά πόσο θα γίνει αποδεκτή η συμφωνία αυτή από το κοινό. Μιλάτε για το σεβασμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών. Φυσικά και συμφωνώ, βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής και θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε αυτές τις πολιτικές. Μιλώ τώρα εδώ ως δικηγόρος γαλλική ένωμη του γραπτού δικαίου και της ε, δυνατότητας του δικαστή να επέμβει ε, είναι κάπως αντιφατικό με αυτές, αυτούς τους κανόνες τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς που είναι πάνω από το 40% της συνολικής συμφωνίας TTIP. Είναι δύνατον ε, να δεχτούμε ότι αυτοί οι κανόνες θα εκφύγουν ε, της δικαιοδοσίας μιας ανεξάρτητης δικαστικής αρχής. Τώρα, για το ISDS ε, δεν είναι θέμα ιδεολογικό, αλλά είτε βρισκόμαστε στη, στα πλαίσια της αμερικανικής λογικής, ε, ε, της διαιτησίας, που κάποιος μπορεί από δικηγόρος να γίνει δικαστή σε διαιτητικό δικαστήριο, αυτή η λογική είναι ασύμβατη με το δική μας νομική παράδοση και ένομη τάξη. Πέραν τούτου θα συνεχίσουμε την διαπραγμάτευση μαζί μας για να βρούμε μια χρήση τομή. Προς το παρόν πάντως οι προτάσεις για το ISDS δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Και ο κύριος Καστάλντι απουσιάζει. Οπότε περνάμε στην κυρία Μάιτε Ρουίς. Ευχαριστώ. Απουσιάζει ο κύριος Γκέρερς, αλλά θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πόνς για την προσπάθειά του. Άρτια και αντικειμενική η γνωμοδότησή του βάζει τις σωστές βάσεις και θέτει τα σωστά ζητήματα. Θα υποβάλουμε βέβαια κάποιες τροπολογίες, ε, αλλά συμφωνούμε και με το υποχρεωτικό Μητρό Διαφάνειας και με την ανάμειξη των Εθνικών Κοινοβουλίων και με διάφορα άλλα θέματα. Θα υποβάλουμε τροπολογίες για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών κράτους επενδυτή, γιατί εκεί έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά εκτιμούμε ιδιαίτερα στην προσπάθειά σας και σίγουρα σε καμία περίπτωση θα πρέπει να παραβιάζουμε το δημόσιο δίκαιο ε, και την δυνατότητα πρόσβασης σε κείμενα που μπορεί να έχουν προσωρινά χαρακτηριστεί ως απόρριτα, αλλά κάποια στιγμή μπορούν να αποχαρακτηριστούν και να χάσουν αυτή τη ε, διαβάθμιση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το δικαίωμα διαφάνειας και πρόσβαση του κοινού θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Πολύ ενδιαφέρουσα πάντω η γνωμοδότηση και συγχαρητήρια για το έργο σας. Παρόλο που θα υποβάλουμε τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ο Αντρέι Πλέγκοβιτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε για την έκθεση αυτή η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ακριβής ε, και μας δείχνει τι μας αφορά ως ε, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και ειδικά όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Συμφωνία TTIP και το Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών όπου κάποιες ε, ανησυχίες έχουν εκφραστεί από την κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει άρα να καθορίσουμε επακριβώς ε, τους ε, ξένους επενδυτές και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε στην έκθεσή σας. Για την ε, διαφάνεια νομίζω πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για ένα δεσμευτικό μητρό έτσι ώστε όλοι οι φορείς της δημόσιας διαβούλευσης όπως αυτή έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνονται παρκώς. Κατά την άποψή μου, η συμφωνία TTIP έχει στρατηγική σημασία, όχι μόνο για την οικονομία και τις επενδύσεις, αλλά βελτιώνει και τη γεωστρατηγική μας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον 21ο αιώνα. Και θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα μέχρι να περάσει η συμφωνία. Ευχαριστώ, Γκέρολ Θάντερντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με τους ε, προλαλήσαντες ε, πως ε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων να μην ασχολούμαστε με όλα τα ζητήματα και ακριβώς είναι ένα από τα θετικά νομίζω της Επιτροπής μας ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Οπότε συμφωνώ με αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα. και νομίζω πως ε, το έχουμε πει αυτό και στην ΛΥΜΠΕ, δηλαδή να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την υγεία, την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια ή με την πολιτισμική κληρονομιά ως πιθανές εξαιρέσεις. κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει μπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια είναι και προστασία της ε, εθνικής γλώσσας η οποία ακόμα δεν υπάρχει στο κείμενο αυτό πουθενά, αλλά για τα υπόλοιπα νομίζω πως μπορώ να συμφωνήσω λίγο πολύ με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελμαρ Μπρόκ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πρόταση. Είναι πάρα πολύ καλή η πρότασή της και ελπίζω να γράψει μια καλή έκθεση. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση γενικότερη. Συνολικά το ελεύθερο εμπόριο είναι κάτι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κατά κανόνα έχουμε εμπορικό πλεόνασμα απέναντι και σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και το να παραμερίσουμε τους μη δασμολογικούς αλλά και τους δασμολογικούς φραγμούς θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. γιατί συνήθως συζητάμε ότι κάτι είναι επικίνδυνο, δεν επιτρέπεται να το κάνουμε κτλ. Και ε, ίσως δημιουργείται μια λανθασμένη εντύπωση για τη γενικότερη αξιολόγηση όσον αφορά την διαφάνεια. Ε, πράγματι δεν ε, γίνεται όμως να κάνουμε τη διαπραγμάτευση στην αγορά. Άμα πάμε και τα έχει διαβάσει στην εφημερίδα ο συνομιλητής μας έχουμε ήδη χάσει στην ε, διαπραγμάτευση σημαντικός πράγματι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, αλλά βεβαίω έχουμε και ένα σώμα ε, των λεγόμενων ενδιαφερομένων διαφόρων ε, οργανώσεων ε, από περιβαλλοντικές οργανώσεις μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε οι οποίες ενημερώνονται πριν από την Κομισιόν. Δεν είναι πάρα Πρέπει να βελτιωθεί εδώ πέρα η κατάσταση. Επίση, τα εθνικά κοινοβούλια δεν είναι δική μα υπόθεση να ενημερωθούν από τι κυβερνήσει που ξέρουν πώ πάνε οι διαπραγματεύσει. Αυτό είναι δουλειά των κυβερνήσεων, όχι δική μα. Και είναι και θέμα αρχής νομίζω, έτσι ο καθένας έχει τις δικές του αρμοδιότητες. Κάτι άλλο σημαντικό επίσης μετά την απόφαση του δικαστηρίου, τη λεγόμενη υπόθεση Φιλιππίνη, κατά πόσον πρόκειται για μία μεικτή συμφωνία ή μία συμφωνία η οποία βασίζεται σε αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πρέπει δηλαδή να κυριωθεί μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή και στις 28 χώρες και φτάνουμε στα 40 ε, κοινοβούλια. Ήδη έχουμε αρκετά κοινοβούλια στο Περολίνο. Και αντιλαμβάνεστε πως ε, τελικά αυτό το ζήτημα του ορισμού μεικτών και μη συμφωνιών είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την διαδικασία της ε, Υπάρχουν 130-140 περιπτώσεις ε, και αφορούν γύρω στους 70 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αλλά αφορά ε, διακριτική ε, μεταχείριση και δεν έχουν ούτε μία επίδραση σε νομοθετικές αρμοδιότητες οι οποίες θα εξακολουθήσουν να είναι τελείως ελεύθερες όπως και αυτές του Αμερικανικού Κογκρέσου οι οποίοι νομίζω έχουν κάθε διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ μας. Μην έχετε την εντύπωση δηλαδή όπως παρουσιάζεται δημοσίως, πως ε, τα κοινοβούλια τα οποία θα το κυρώσουν έχουν κάποια διάθεση να δώσουν τις αρμοδιότητές τους σε κάποιο σώμα διαιτησίας. Και πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα στην σύνταξη ήδη της ε, συνθήκης. Αλλά είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις, μάλλον πω το εξή. Αν νομοθετήσουμε εμείς στην Ευρώπη για το περιβάλλον, η νομοθεσία αφορά εξίσου ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες. Και δεν είναι δυνατόν βεβαίω να επιβαρύνει μόνο τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Αυτό είναι το θέμα. Και μην ξεχνάμε πως οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Αμερική είναι μεγαλύτερες από ό,τι οι αμερικανικές στην Ευρώπη. Μόνο και από αυτό μας συμφέρει. Γιατί εάν πάμε στα εθνικά δικαστήρια εξαρτώμαστε από την ομοθεσία της κάθε χώρας την οποία καθορίζει η κυβέρνηση. Οπότε αν κάποιος υφίσταται διακριτική μεταχείριση θα χάσει και στο δικαστήριο. Και βεβαίω ε, ούτω ή άλλω, ε, το να μπει στη δικαστική διαδικασία στη ΣΥΠΑ με το τεράστιο κόστος σημαίνει πως έχει χάσει ούτω ή άλλω εξ αρχής. Οπότε εδώ πέρα ε, να περιοριστούμε στο θέμα της διακριτικής μεταχείρισης ή όχι και να τελειώσει εκεί. για να εγκριθεί και η συνθήκη. Και να πω κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να το πούμε περισσότερο δημοσίως. Στην δημόσια συζήτηση δεν είναι γνωστό ότι η συνθήκη αυτή, όπως κάθε εμπορική συνθήκη, κυρώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχει ήδη αποτελέσει ε, αντικείμενο διαπραγματεύσεων. και έχουν γίνει ήδη ακροάσεις ε, και στο κοινοβούλιο όλα αυτά. Αυτά πρέπει να τα παρουσιάσουμε, να μην έχει το κοινό την εντύπωση πως πήγε η Κομισιόν και διαπραγματεύτηκε κάτι στα κρυφά και αυτό ήταν. Αυτό δεν μας απασχολεί εδώ και χρόνια αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ πάλι, Ράντσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και εγώ τον Στέβαν ε, Γκονσάλες Πόνς. Είναι μια πολύ ισορροπημένη τοποθέτηση. Η μόνη ανησυχία που θα έχω καθότι έχει εκφραστεί σε διάφορα εθνικά βήματα είναι αυτή η επίλυση των διαφορών συμφωνώ με τον Έλμαρ ότι μάλλον η σύγκρουση δεν είναι νομοθετικής φύσεως αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια απώλεια εμπιστοσύνης στα δικαστήρια και στην κοινή γνώμη. Υπάρχει ένας φόβος δηλαδή ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα αυτά ώστε να επιβάλλουν κάποιους διαφοροποιημένους, κάποιους διαφορετικούς κανόνες διαιτησίας. Και ίσως να είναι λίγο φιλόδοξο, αλλά έχουμε ένα σύστημα που θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε περαιτέρω, ώστε να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα μόνιμο φορέα επίλυσης διαφορών και όχι κατά περίπτωση να τον δημιουργούμε. Ώστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρχει μια τέτοια θεσμική επιλογή και θεσμική εγγύηση σχετικά με την οποιαδήποτε επίλυση. Και για την επιλογή των μελών ενός τέτοιου δικαστηρίου φορέα θα έπρεπε να, να συσχετίζονται θεσμικός πώς και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή οι δύο όχθες του Ατλαντικού. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικά φιλόδοξη η πρότασή μου. Ε, ε. Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εφικτή. Γιατί υπάρχουν διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι εν εξελίξη αλλά ίσως να είναι μια ενδιάμεση λύση. Όχι η απόλυτη καθαρή λύση διαιτησίας που δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε να είναι υπερβολικά άκαμπτη. Γιατί χρειαζόμαστε συχνά ταχύες αποφάσεις ανεξαρτήτως από τα εθνικά σώματα, από τους εθνικούς φορείς. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα σκεφτώ, θα εξετάσω μια τροπολογία που θα μπορούσα να σας προτείνω, να σας υποβάλω προς την κατένιση αυτήν, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε έναν μόνιμο φορέα, ένα μόνιμο δικαστήριο επίλυση διαφορών. Ήδη στη Χάγη έχουμε κάτι τέτοιο. Και ένα τέτοιο θεσμικός φορέας θα έδινε εμπιστοσύνη. Ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκούς φορείς, γιατί στην Αμερική έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο σύστημα. Στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες η ίδια αντίληψη. Έχουμε και έναν πρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής αν θέλετε σύντομα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και ε, τους συζητητές. Κάποιες διευθυνήσεις μόνο από πλευράς μου ή τουλάχιστον να προσπαθήσω να σας ε, διαβεβαιώσω. Μιλούμε για ένα συμβούλιο, ένα αριθμιστικό συμβούλιο συνεργασίας δεν μιλούμε για έναν φορέα λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί δεν μπορεί και δεν πρέπει να θέτει ένα αμφιβόλο τη συνταγματική διαδικασία λήψεως απόφασης. Ούτε βεβαίως τις αρμοδιότητες του οίκου σας και οποιοδήποτε άλλου. θα λειτουργεί κατά απολύτως αντίστοιχο τρόπο με εκείνον που λειτουργούν ήδη οι Αμερικανοί και επιπροσθέτως για να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε κάποιες συγκλήσεις αλλά διατηρώντας την επιφύλαξη και την ελευθερία να επιβάλλουμε την προστασία που θέλουμε. Το επίπεδο προστασίας που θέλουμε. Το, για το ISDS, για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών δηλαδή μεταξύ επενδυτών και κρατικών φορέων, έχουμε κάποιες κατακρίσεις οι οποίες έχουν σημειωθεί και προσπαθούμε να τις αποφύγουμε. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν και έχουμε ήδη προτείνει ε, τουλάχιστον στα πλαίσια της συμφωνίας με τον Καναδά είναι ένα εξυγχρονισμένο σύστημα ISDS που δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με εκείνο που βρίσκουμε στις διμερείς ε, συμβάσεις ε, ε, τις επενδυτικές ή τις συμβάσεις συνεργασίας. Προσπαθούμε να έχουμε σαφείς κανόνες ώστε να μην αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες εκτός πλαισίου δηλαδή σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Ντιόν ε, στην ΣΥΤΑ υπάρχει με τον Καναδά μια σαφής ρήτρα που προβλέπει ότι δεν μπορεί να επικαλούμαστε οποιαδήποτε διάταξη η οποία να υπερβαίνει τα πλαίσια που έχουμε συμφωνήσει διμερός ή πολυμερός ανάλογα με το πώς έχει περιπτώσει, ανάλογα με τη δικαιοδοσία του κάθε δικαστηρίου. Έχουμε και νέους κανόνες δεοντολογίας και ηθικούς κανόνες. Όλα αυτά έχουν εγγραφεί, έχουν ενσωματωθεί στην συμφωνία με τον Καναδά που γενικώ αναγνωρίζεται ότι είναι ένα ε, βήμα προς τα εμπρός. Και πέρα από τις δημόσιες διαβουλεύσεις που είχαμε ε, για το σύστημα ESDS εντός της TTIP, βλέπουμε και επί νέων ιδεών για να εξυγχρονίσουμε το σύστημα αυτό επίλυση διαφορών. Ε, στις 18 Μαρτίου η κυρία Μάλστρομ θα προσέλθει προκειμένου να ε, παρουσιάσει κάποιες πρώτες ιδέες ε, σχετικά με ένα δευτεροβάθμιο δικαστηρίο το οποίο θα μπορούσε, θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει σε ένα πιο θεσμοποιημένο σύστημα επίλυσης διαφορών. Όπως ανέφερε και ο κ. Ραγγέλ, βεβαίως είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, διότι οργανωτικά και χρηματοδοτικά έχει κάποιες επιπτώσεις, αλλά είναι κάτι που προετοιμάζουμε τον εαυτό μας να εξετάσουμε και επί της διαφάνειας την επόμενη εβδομάδα θα απαντήσει στο διαμεσολαβητή, στην έκθεση δηλαδή η Κομισιόν. Αρκετές από τις συστάσεις του διαμεσολαβητή ήδη έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή όλες οι προτάσεις στα πλαίσια της TTIP είναι ήδη δημόσια διαθέσιμες στην ιστοσελίδα για τη ρυθμιστική συνεργασία, τους σχετικούς φορείς, όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα από την περασμένη εβδομάδα και θα καλούσα όλους εσάς να τα δείτε. Να δείτε δηλαδή όλα αυτά τα εμπιστευτικά ή ευαίσθητα εμπάσχετος έγγραφα που μοιραζόμαστε στα πλαίσια της διαμαράντασης αυτής και μπορούν όλοι οι φορείς να λαμβάνουν και αντίγραφο έντυπο. Θα δείτε λοιπόν περισσότερα στην απάντησή μας την ερχόμενη εβδομάδα προ στον διαμεσολαβητή, η οποία εξάλλου θα δημοσιοποιηθεί. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Πον. Πόνς, ευχαριστώ πρόεδρε. Με πάρα πολύ μεγάλη συντομία να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν σε αυτήν την, ε, την γνωμοδότηση γιατί θεωρώ ότι πολύ σωστά θέλουμε αυτή η έκθεση να είναι μια έκθεση που όλοι προσωπικογράφουν και όχι απλώς μια πλειοψηφία της Επιτροπής. Επομένως καλοδεχούμενες θα είναι όλες οι τροπολογίες και όλες οι παρατηρήσεις ώστε να έχουμε τελικώς μια τοποθέτηση, μια γνωμοδότηση προς την οποία θα συμφωνούν όλοι. Και σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Μπρόκ ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει στην ε, ε, απόφαση και θα πρέπει να υπερασπιστεί των συμφερόντων πολιτών. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι μια μεικτή συμφωνία και ότι θα μπορούσαμε να πάμε πολύ μακριά και να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που κάποιο εθνικό κοινοβούλιο δεν θα επικυρώνε. Πρέπει δηλαδή να συμμετάσχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Και για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών αυτός ήταν εκεί, δεν τον φανταστήκαμε εμείς, δεν τον επινοήσαμε εμείς. Είναι καλύτερα να μιλούμε για αυτόν, γιατί τον έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Εμείς βεβαίως δεν είμαστε το σώμα το οποίο διαπραγματεύεται και επομένως δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να συζητήσει σχετικά με αυτό. Αυτό που μας αντιστοιχεί είναι να πούμε ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός και όχι ποιος θα είναι. Πρέπει να θέσουμε τις κόκκινες γραμμές που δεν μπορεί να ξεπερνάει ο μηχανισμός αυτός και επομένως σχετικά με το θεσμικό όριο που θα πρέπει να σέβεται ο μηχανισμός αυτός νομίζω ότι είναι αρκετά απλό, εν πάση περιπτώσει πραγματοποιήσιμο να συμφωνήσουμε. Ο κύριος Άντρισεν ήθελε ακόμα να μιλήσει ε, για την τύπη, γιατί είχαμε μόλις ε, ολοκληρώσει αυτό το ζήτημα, αν είναι πολύ σημαντικό. Α. Γιατί έχουμε και την ε, προθεσμία, που είναι αρκετά γενναιόδορη, 5 Μαρτίου, θα υπάρχει υπαρκής χρόνος πιστεύω να υποβληθούν, να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Και θα ήθελα να κλείσω αυτό το ζήτημα. 5 Μαρτίου λοιπόν η προθεσμία για τις τροπολογίες μεσημέρι, δεν ξέρω τι έχουμε πει, γιατί εδώ δεν λέει κάτι. Το απόγευμα, 6 ε, ώρα, αφού δεν, δεν λέμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Αποφασίζουμε πολιτικά, εφόσον δεν μας είπατε πιο τεχνικά. Ε, λοιπόν, τώρα ε, θα αναβάλουμε το σημείο 11 για την ε, Γιούρη. Δεν έχουμε χρόνο. Για το 10 ε, θα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Ο κύριος Γεζόφσκι ήταν πολύ... Είχε όλη τη διαθεσιμότητα να δώσει την εισαγωγή, αλλά θα έχουμε τη συζήτηση την επόμενη φορά. Αλλά μπορούμε εδώ να ξεκονομήσουμε ήδη κάποιο χρόνο. Ο κύριος Γεζόφσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για γνωμοδότηση της, Επιτροπή μας, ε, της Επιτροπής μας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, για την εφαρμογή της ε, Αρχής Επικορικότητας και Αναλογικότητας και τις αιτήσεις σχετικές εκθέσεις 2012-2013. Η γνωμοδότηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Επιδοκιμάζει η γνωμοδότηση το γεγονός ότι η Επιτροπή ελέγχει εκ των προτέρων εάν οι προτάσεις της είναι απαραίτητες και αν οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη-μέλη, δηλαδή την αρχή της επικουρικότητας. Επίσης, υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα Εθνικά Κοινοβούλια και προτείνει και τρεις συστάσεις ε, για παράδειγμα την παράταση της προθεσμίας των 8 εβδομάδων που διαθέτουν τα Εθνικά Κοινοβούλια για να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη, προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο ε, για να ενημερωθούν για το θέμα και να συμμετέχουν πιο ενεργά στο διάλογο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Επίσης ε, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει πιο ουσιαστικά κριτήρια για τη διαπίστωση της παραβίασης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, γιατί δυστυχώς ε, δεν υπάρχει συνοχή στον τρόπο ερμηνείας ε, των αρχών αυτών από τα κράτη-μέλη. Αυτό μας έχουν υποδείξει πολλοί εμπειρογνώμονες. Και τέλος ε, παρατρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει με ευνοϊκότερο και πιο ανοιχτό τρόπο την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να επηρεάζουν περισσότερο την ενωσιακή νομοθεσία. Αυτά νομίζω ότι επικεντρώθηκα στα ουσιώδη και χωρίς να μακρηγορώ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση θα γίνει στην επόμενη μας συνεδρίαση γιατί θέλαμε να απελευθερώσουμε λίγο χρόνο μια και στι 6 ε, παρατέταρτο θα έρθουν οι συνάδελφοι τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την κοινή μα συνεδρίαση. Θα παρατείνουμε αντίστοιχα και την διορία για την ε, κατάθεση των τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μα στις 16 Απριλίου, οπότε χρόνο έχουμε. Το σημείο 11 το αφήνουμε και επανερχόμαστε στα σημεία 7 και 8. Έχουμε μία ώρα για τη συζήτηση των δύο εκθέσεων. Και θα ήθελα να μας κάνετε την εισαγωγή μια ναι, και δεν έχετε έτοιμα έγγραφα, αλλά θα ήθελα να μας παρουσιάσετε τις απόψεις για να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε. Έχουμε μία έκθεση ε, με εισηγητές, συνεισηγητές, τον κύριο Μπρό και την κυρία Μπρέσο και μία έκθεση του κυρίου Φερχόφστατ που λέει τι γίνεται μετά τη συνθήκη. Δεν ξέρω ποιος ε, θα πάρει πρώτα στο λόγο. Κυρία Μπρέσο. I can start. prima, ε, di tutto ε, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με μία εκτίμηση που κάναμε μαζί με τον συνάδελφο Μπρόκ και τον συνάδελφο Βερχόφστατ. Δηλαδή, να έχουμε ένα κοινό εισαγωγικό σημείωμα και για τις δύο γνωμοδοτήσεις που να καθορίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση και που να εξηγεί ότι κάποιες από αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μιας εντελεχέστερης εξέτασης των συνθήκων, ενώ άλλες θα απαιτούσαν τροποποίηση των συνδικών. Δηλαδή κατά πόσον θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένα μέσο μιας νέας συνέλευσης ή οποιαδήποτε άλλο μέσο που θα μπορούσε να προσφέρει η συνθήκη. Ε, εν ολίγης τις νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου που, τις οποίες δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει πλέον αυτά τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθότι θεωρούσαμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θεωρούσαμε ότι θα είχε μπροστά της ε, λούσια όπως είναι η συνθήκη αυτή ένα μεγάλο διάστημα χρονικό. Οι θεματικές είναι βασικώς δύο. Καταρχάς η χρηματοπιστωτική κρίση η οποία δοκιμάζει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση την ίδια και έχει καταδείξει τα όρια αντοχής, θα έλεγε κανείς, τη συνθήκη στο πεδίο αυτό. Γνωρίζετε ότι απέναντι στην κρίση αυτή αρκετές χώρες χρειάστηκε να βρουν λύσεις ζορίζοντας λίγο τα όρια των συνθήκων, αλλά και μέσω συμβάσεων πρόσθετων, που θα πρέπει να συμπεριληφθούν, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη συνθήκη. Τώρα, άλλο, άλλη μια θεματική, ακόμα πιο πρόσφατη, δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο διεθνές επίπεδο, στη διεθνή σκηνή. την κατάσταση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, την επίκουσα κατάσταση απέναντι στον Ισλαμικό φονταμεταλισμό το οποίο καταδεικνύει ότι λείπει μία συνεπής και κοινή εξωτερική γραμμή και πολιτική. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ε, σημειώσαμε, είδαμε μια ε, ηγετική στάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μέσω και της πρωτοβουλίας των τεσσάρων προέδρων έχει θέσει ε, ένα πλαίσιο προκλήσεων που εντός των οποίων πάντοτε ελοχεύει το θέμα της πολιτικής ένωσης. Και τελικά δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποια αποτελέσματα επιτεύχθησαν, αλλά χρειάζεται μια νέα οικονομική διακυβέρνηση και χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε με τα υφιστάμενα μέσα αλλά και με πρόσθετα μέσα τα θέματα της ασφάλειας των, της πολιτικής άμυνας της πολιτικής της εξωτερικής και υπάρχει και ένα ζήτημα δημοκρατικότητος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραγωνίστηκε θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών από κάποιες ε, επίγουσες καταστάσεις χρησιμοποίησε θετικά βεβαίως τη συνθήκη της Λισαβόνας προκειμένου να εκλέξει δημοκρατικά τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα σύστημα που είναι πολύ ενδιαφέρον διότι αυτό ενισχύει τις πολιτικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά για το μέλλον θα χρειαστεί μια πληρέστερη εξέταση του πώς η δημοκρατική νομιμοποίηση της επιλογής των επιτρόπων και της Κομισιόν θα μπορούσε να ενισχυθεί. Ήδη αναφέρθηκα ε, στους τέσσερις πρόεδρους προκειμένου να πάμε σε μια αυθεντική οικονομική και νομισματική ένωση ο στόχος θα έπρεπε να είναι εκείνος μιας πιο ολοκληρωμένης πολιτικής ένωσης. Και η τελευταία έκθεση που προετοιμάζουν οι τέσσερις πρόεδροι κάνει κάποια δειλά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, το οποίο καταδεικνύει ότι είμαστε σε μια οριακή κατάσταση. Δηλαδή έχουμε μέσα εντός της ε, υφιστάμενης συνθήκης που μας επιτρέπουν να πάνε προς μια κατεύθυνση πιο ολοκληρωμένης ε, ενώσης εφόσον τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι θεσμικοί φορείς το επιθυμούν αλλά έχουμε και τη δυνατότητα ενδεχομένως να έχουμε διαφορετικών εναλλακτικών ε, συστημάτων ή πλαισίων που να βελτιώνουν τη δημοκρατικότητα του συνόλου. Ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η οικονομική και ιδιαίτερα η νομισματική κρίση της Ευρωζώνης απαιτεί μια αποτελεσματική πολιτική οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπό την έννοια αυτή όλες οι προτάσεις που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων για την επιλογή του Προέδρου της Κομισιόν καταδεικνύουν ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο στενή, πιο ολοκληρωμένη ένωση. Προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και όχι μόνο της νομισματικής. και έγιναν πάρα πολλά, διαδέχθηκαν επεισόδια το ένα το άλλο, ε, σύνοδοι κορυφής, ευρωπαϊκά συμβούλια, ε. και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε την κατάσταση επαναλαμβάνω εντός του πλαισίου των υφισταμένων συνδικών αλλά ίσως και με νέα στοιχεία νέα συνταγματικά εν περιπτώσει στοιχεία Ακινούμε λοιπόν από μια, ένα κοινό πυρήνα εξέτασης, ανάλυσης ε, προβλημάτων και από εκεί και πέρα ε, σε ό,τι μας αφορά θα είναι το κατά πόσον ε, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια πιο διαφανή, πιο δημοκρατική κοινή ε, οικονομική πολιτική, κοινή πολιτική άμυνας, ενέργειας, ε, ε, χρηματαγορών, δηλαδή όλων εκείνων των στοιχείων που αρκετές εκθέσεις των τεσσάρων προέδρων καθόρισαν αλλά επί των οποίων δεν έχει ακόμα μπει μια τάξη και θα έκλεινα λέγοντας το εξής, ακόμα και η χρησιμοποίηση του όρου ένωση χρειάζεται κάποια θεσμική διευκρίνηση. Το βλέπουμε συνεχώς. Μιλούμε για την Τραπεζική Ένωση, την Ενεργειακή Ένωση, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ποια είναι η θεσμική δομή αυτής της Ένωσης ή αυτών των ενώσεων επί παραδείγματι. Μιλούμε για έναν πρώτο, έναν αρχικό πυρήνα, ένα πρώτο βήμα κάποιων αρμοδιοτήτων τον, τους, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική στην οποία προσθέτουμε εθελοντικές δεσμεύσεις των κρατών αλλά μια εθελοντική εκχώρηση, δέσμευση των χωρών δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο όρος ένωση υποκρύπτει πολύ διαφορετικά πράγματα. Ένα παλίμψιστο από πολιτικές ή ένας κοινός προσανατολισμός καλά ορισμένος και εν πάση περιπτώσει δεσμευτικό. Νομίζω ότι και η δική μας Επιτροπή εδώ θα πρέπει να επιχειρήσει να με σαφήνεια να διευκρινίσει τι εννοούμε όταν λέμε ένωση. Και όταν μιλούμε για ένωση χ ή Ψη αμήνης ενεργείας τραπεζική, να το ορίζουμε αυτό καλύτερα θυσμικός, δηλαδή συνταγματικός πώς. Η ιδέα έκθεση του Βερχόφσταντ είναι συνδεδεμένη γιατί εφόσον αποφασίσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση του θεσμικού πλαισίου θα πρέπει να, τελικά να εξετάσουμε μια δεχόμενη τροποποίηση. Θεσμική μεταρρύθμιση. Το οποίο δεν μπορεί παρά να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πρωταγωνιστή. Έχουμε τη δομή της συνέλευσης που θα μπορούσε να ζητήσει το Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε και αυτός είναι ακριβώς ο σχετισμός μεταξύ των, της μίας και της άλλης εκθέσεως. Δηλαδή, μία από τις εξουσίες, της αρμοδιότητες που δεν έχει χρησιμοποιήσει το Κοινοβούλιο είναι η εκκίνηση μιας νέας συνέλευσης. Αλλά αυτό θα σήμαινε ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι δεν έχει επαρκείς αρμοδιότητες η Ένωση σε κάποια πεδία και ότι θα έπρεπε να οριστούν, να τροποποιηθούν να συμπληρωθούν ή και να υπάρξουν αφαιρέσεις. Δεν μιλάω μόνο με θετικό πρόσημο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλμαρ Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Αν και επί της ουσίας συμφωνώ με την κυρία συνάδελφο. Φαίνεται πως σημαντικό είναι το ότι οι τρεις ε, εισηγητές βλέπουν την, ε, τις εκθέσεις τους ως μια ενότητα με διαφορετικούς στόχους. Η κυρία Μπρέσο και εγώ να ζητούμε δυνατότητες για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την συνθήκη της ε, Λισαβόνας σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο. Ο Γκί εντωμεταξύ βεβαίως ε, έχει ένα όραμα για το μέλλον. Αλλά όλα αυτά εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο. Και βεβαίω έχει σημασία η διαδικασία λήψη ε, αποφάσεων. Αυτά τα οποία λέει η κυρία Μπρέσο πρέπει να τα εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Είναι μια δουλειά αυτή την οποία κάνει ο Γκίφερ Χόφστατ έτσι ώστε αν καταλήξουμε στην επόμενη ε, συνταγματική συνέλευση να είμαστε έτοιμοι. Αυτό σχετίζεται και με τη συζήτηση για τη Μεγάλη Βρετανία και για την ΟΝΕ. Και έτσι μπορεί, γιατί κοιτάξτε, μπορεί να έχουμε εξελίξεις και να βρεθούμε ξαφνικά γρήγορα μπροστά σε ε, συζητήσεις για αλλαγή τη συνθήκης. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα συγκεκριμένα και κάποια άλλα πιο γενικά. Το ένα, Κοιτάξτε, εντός ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόμαστε μονίμως σε μία ρευστή, δηλαδή μπορούμε να λειτουργούμε και με την αρχή ε, του Δελόρ, παραδείγματος χάρη στην ΟΝΕ και να κινούμαστε αρκετά γρήγορα και αυτό σημαίνει βεβαίως πως δεν θα πρέπει ποτέ να έχουμε θεσμικά κενά, χάσματα. Και ουσιαστικά και γραφειοκρατικά και κενό παραδείγματος χάρη μεταξύ ε, χωρών ε, της ζώνης ευρώ και των λοιπών. Η Κομισιόν, παραδείγματο χάρη, είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη Κομισιόν για την Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλος πρόεδρος του Eurogroup θεσμικά μιλώντας, είναι ενιαία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω ε, όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση στην ΟΝΕ θα πρέπει αυτή πάντα να μην οδηγεί αυτό το λανθασμένο συμπέρασμα το οποίο μόλις περιέγραψα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λογική απάντηση που θα διατηρεί αυτή την νότη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μας δίνει δυνατότητα βίως να μπορούμε να κινηθούμε και να δράσουμε. Εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα του τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δρά πάντα ενιαίο ή μπορεί να κινητοποιηθεί ένα τμήμα του μόνο αυτό θα έχει σοβαρές, ε, σοβαρότατες ε, συνέπειες ε, στον τομέα της δημοκρατίας. Εγώ για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση είμαι πάντα υπέρ των ενιαίων και συνολικών λύσεων. Όπως είπα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δρούμε στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και βεβαίως εδώ πέρα πηγαίνει και η έκθεση Γκουλάρ. Και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη για να δούμε σε τι τελικό αποτέλεσμα θα καταλήξουμε, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες, ε, τι γίνεται με εθνικό και ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Δεν χρειάζεται νομίζω να συνεχίσω. Να συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το πλαίσιο εκείνο που σχετίζεται με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας. Τι γίνεται μεταξύ των θεσμικών οργάνων, τι κάνουμε με την μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και με άλλα ζητήματα όπου πρέπει να είμαστε σε δυνατότητα να λειτουργούμε γρήγορα. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της συνολικής ε, χρηματοδότησης της ε, εξωτερικής ε, πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Η αρχή αυτή που υπάρχει ήδη πρόκειται για ένα σχετικά νέο τομέα και θα πρέπει να δούμε και εδώ πέρα ποια είναι τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να τα συζητήσουμε. Έχουμε λοιπόν και τα κλασικά ζητήματα. δείτε τι γίνεται με το άρθρο 20 και το και το άρθρο 126 της συνθήκης, τη λεγόμενη ενισχυμένη συνεργασία. Τι θα γίνει με τα νέα δικαιώματα ε, ψήφου του Κοινοβουλίου και τη συμμετοχή στο Συμβούλιο μέχρι το 2017. Επίσης, πάρα πολύ ενδιαφέρον τι θα γίνει με τις ε, ρήτρες αυτές, ε, τις λεγόμενες ε, πασαρέλες ε, ε, με τις οποίες ε, σκοπεύουμε να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργεί. Ξέρω πως απαιτείται ομοφωνία, αλλά είναι ένας τρόπος τουλάχιστον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Και αυτό βέβαια αφορά την ΟΝΕ. Και νομίζω πως το θέμα το οποίο σχετίζεται με το άρθρο 136 ε, έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα μου αλλά δεν το αντιλαμβάνεται αυτό η Γερμανία ε, υπάρχουν φοβισμένοι δικαστές στην ε, Καλσρούη και ζητάνε νομικές διαβεβαιώσεις για το ότι δεν μπορεί να παραβιαστεί αυτό το άρθρο και εάν υπήρχαν πραγματικά αυτές οι διαβεβαιώσεις ε, νομίζω θα μπορούσαμε και εμείς να κινηθούμε πάρα πολύ πιο άνετα και να περάσουμε άλλα πράγματα μέσα στην συνθήκη παραδείγματο χάρη την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να κινείται ανεξάρτητα. Πάλα πολλά πράγματα πράγματι γίνονται από τον φόβο του Εθνικού ε, Συνταγματικού Δικαστή και για να τα αποφύγουμε αυτό πηγαίνουμε συνεχώς σε ένα διακυβερνητικό πλαίσιο. Βεβαίω έχουμε συμφωνήσει πως μέσα σε πέντε χρόνια θα πρέπει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο να μπει στην συνθήκη. Πρέπει να αρχίσουμε γιατί τα πέντε χρόνια περνάνε γρήγορα και υπάρχουν οι υποχρεώσεις του Προέδρου του Eurogroup, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του τότε Επιτρόπου Νομισματικών που έχουν αναλυφθεί για αυτά τα ζητήματα. Είχαμε ανταλλάξει τότε επιστολές, ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ ήταν τότε στην άλλη πλευρά και με βοήθησε και διαπιστώσαμε πως αυτός είναι ο στόχος. Έτσι δώσαμε και την ε, σύμφωνη γνώμη μας. Και έτσι θα πρέπει νομίζω να ε, προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Κυρίε και κύριοι, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Π.χ. τι θα γίνει με το βρετανικό θέμα. Χθε είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Βρετανό Υφυπουργό ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και να συζητήσουμε βεβαίω το θέμα των αρμοδιοτήτων και πώς μπορεί να καθοριστεί πολιτικά για να μην χρειάζεται αλλαγή η συνθήκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω αυτό. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ως κοινοβούλιο πως καλοί μας άνθρωποι δεν χρειάζεται να αλλάξει συνθήκη για αυτό το οποίο ζητάτε. Είναι απλό, γίνεται χωρίς αλλαγή. Τότε είναι σημαντικό αυτό το θέμα και εδώ πέρα βεβαίως ε, υπάρχει και το άλλο θέμα που προκύπτει από τη Βρετανία τα δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας. Ε, Εμεί ως Κοινοβούλιο στι διαπραγματεύσεις με την Ολλανδία η οποία έχει απορρίψει την συνταγματική συνθήκη την ε, προηγουμένη της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, είχαμε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό Μπάλκενέντε ο οποίος συζήτησε να μπει μια ε, ρήτρα για τα δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων, η οποία όμως ε, δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. Είναι σαφές πώς. Όταν ε, κάποιο κοινοβούλιο είναι εναντίον ε, της νομοθεσίας ε, είτε λόγω μονομερών ε, ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε του Συμβουλίου έχει τελειώσει εκεί πέρα η υπόθεση. Τα Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε βέβαια να τους δώσουμε ε, τη δυνατότητα να είναι, αν θέλετε, ένα τρίτο νομοθετικό σώμα, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εμπιστοσύνη, μια σχέση εμπιστοσύνης με τα Εθνικά Κοινοβούλια, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια αλλαγή των αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της συνθήκης. Η κυρία Αγκουλάρ τώρα πρότεινε κάτι που το οποίο δεν μου αρέσει. Όταν μιλάμε για μικτές αρμοδιότητες, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είτε είναι εθνική αρμοδιότητα, είτε ευρωπαϊκή και έχει το ανάλογο κοινοβούλιο την ευθύνη. Όχι και τα δύο όμως, τότε δεν είναι κανείς υπεύθυνο. Διευκρινήσει, ναι, αυτό νομίζω μπορούμε να το κάνουμε, έχει γίνει πάρα πολλέ ε, φορές. Αυτά άλλα πράγματα. Έχουμε ε, και το καθεστώς των ε, κομμάτων. Αναφέρονται στην ε, συνθήκη, έχουν ένα αλλά θα πρέπει να δούμε και την σημασία των πολιτικών κομμάτων. Και είναι σημαντικό αυτό για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. όσο δεν έχουμε ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία θα κατεβάζουν ε, τις λίστες εγκαίρως πριν από τις ε, ευρωεκλογές ε, δεν θα ισχυροποιηθεί ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι μονίμως αντικείμενο πίεσης και συμβασμών και έχουμε ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα εκεί πέρα και βεβαίως έχουμε και το αγαπημένο μου θέμα εγώ θα ήθελα να γίνει κάποιο είδους ε, άνω βουλή το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αναφέρεται, όχι τα Συμβουλία στην συνθήκη και εγώ θα ήθελα να συνεδριάζει δύο-τρεις φορές το μήνα ως κάποιο είδους ε, άνω σώμα, σε ανοιχτή συνεδρίαση δηλαδή, να το βλέπουν όλοι για τα για το νομοθετικό όργο Και τα Υπουργικά Συμβουλία να γίνουν επιτροπές του Συμβουλίου. Τα Συμβούλια Υπουργών και από μια τέτοια ανοιχτή συζήτηση δημόσια να προκύψει η διαφάνεια την οποία χρειαζόμαστε. Και αυτό σημαίνει βεβαίως πως εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να φύγουμε τελείως από την ε, πρώτη ανάγνωση. Η φυσιολογική νομοθετική διαδικασία πρέπει να περιέχει δύο αναγνώσεις. Αυτές οι συμφωνίες στην πρώτη ανάγνωση και βγαίνει από θέση ισχύω ε, ο εισηγητής ε, και τα συζητάει με τον πρέσβη δεν είναι τρόπος αυτός να γράφουμε νόμους δεν είναι δημοκρατική νομοθετική διαδικασία. Σε ένα κλασικό νομοθετικό σώμα σε περισσότερα εθνικά κοινοβούλια γίνονται τρεις αναγνώσεις και μεταξύ αυτών των αναγνώσεων μπορούν να επηρεάσουν οι ενδιαφερόμενοι να γίνει μια δημόσια συζήτηση και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσουν την νομοθεσία. Είναι σημαντικό αυτό για την αξιοπιστία της νομοθεσίας μας, γιατί κάνουμε από ένα τριμερή διάλογο, εμφανίζεται ένας νόμος και απορρίξει ξαφνικά ο πολίτης ότι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ αντιλαμβάνομαι τους πολίτες όταν δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος γιατί και πότε. Και βεβαίω όταν δεν το καταλαβαίνει κανείς είναι εναντίον. Η ίδια συζήτηση με το TTIP. Και ελπίζω πραγματικά να ε, ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα όπως επίσης και η διαδικασία της διαμεσολάβησης το οποίο από πλευράς δημοκρατίας είναι κάτι το φεδρό εμείς είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε συγητές και πόση εξουσία έχουμε αλλά δεν είναι λογική αυτή πρέπει λοιπόν εδώ πέρα πραγματικά να αναρωτηθούμε αν θα παίξουμε αυτόν τον... αν θέλουμε να παίζουμε αυτό το ρόλο. Είχα και κάτι άλλο τώρα, το ξέχασα νομίζω φτάνει με αυτά. Α, μια διαπίστωση. Πρώτα απ' όλα, ο πρόεδρος του Eurogroup σύμφωνα με τη συνθήκη μπορεί να είναι και ο επίτροπος ο αρμόδιος για τα νομισματικά. Έτσι θα λυθούν κάποια πραγματάκια, κάποια προβληματάκια. Και κάτι άλλο. μπορεί ο πρόεδρος της Κομισιόν ταυτόχρονα να είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρέπει να θυμηθούμε πως υπάρχουν αυτές οι ε, δυνατότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Ευχαριστώ. Και πάμε κατευθείαν ε, σε εσά και κατόπιν θα γίνει κοινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, για τη μεθοδολογία που ακολούθησαν η κυρία Μπρέσο και ο κύριος Μπρόκ. Θα καταλήξουμε σε ένα κοινό έγγραφο εργασία ε, ε, με μία νέα ανάλυση, γιατί θα ήταν ανόητο να έχουμε δύο διαφορετικές εκθέσεις και δύο διαφορετικές αναλύσεις για το ίδιο θέμα. Κάτι βέβαια ε, δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα συνέβαινε στην πολιτική, αλλά Προσπαθούμε να το αποβίγουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά. Να έχουμε μία ενιαία, μία κοινή ανάλυση και ένα έγγραφο. Βέβαια το, το θέμα μας είναι διαφορετικό. Μιλούμε για το δυναμικό ε, της συνθήκης και για τις εξελίξεις εκτός της συνθήκης. Αλλά καλό θα ήταν να συντονίσουμε τις ε, θέσεις μας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα να ετοιμάσουμε το έγγραφο εργασίας πριν το καλοκαίρι. Μάιο, Ιούνιο, αυτός είναι ο στόχος. Και να δημιουργήσουμε αυτό το έγγραφο εργασίας, μία βάση, ώστε να έχουμε την πρώτη έκθεση γύρω το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Δεν θα αποφασίσω εγώ ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα ε, του, τις εκθέσεις του κυρίου Μπροκ, αλλά νομίζω θα ήταν καλός αυτός ο χρονικός ορίζοντας. Και η δεύτερη έκθεση αναμένεται για τα τέλη του έτους. Η δεύτερη έκθεση που μιλάει για τις προοπτικές εκτός συνθήκης και μετά τη συνθήκη. Τώρα, τι γίνεται με τη δεύτερη έκθεση, πώς θα την προσεγγίσουμε. Θα εφαρμόσουμε αυτά που έγιναν το 53, το 67, το 2001, το 2005 που ήταν όλα ανοιχτά γιατί είπαμε θα συγκαλέσουμε συντακτική συνέλευση που στηρίχτηκε στη διακήρυξη του Λάκεν αλλά είχαμε και προηγούμενες απόπειρες το 53 το είχα ξεχάσει τελείως τώρα μου ξαναήρθε σίγουρα θα έχουμε πολλά παραρτήματα και το 67 μία από τα ίδια ήταν ανοιχτά όμως τα πάντα. Λέμε να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα θεσμικό σύστημα. Το 53 δεν είχαμε σχεδόν τίποτα. Και η συνέλευση το 2001-2005 επίσης είχε σχετικά ανοιχτή εντολή. Ξεκίνησε σχεδόν εκ του μηδενός. Τεράστιες ευκαιρίες δηλαδή και δυναμικό. και οι δύο άλλοι εισηγητές συμφωνούν να μην επαναλάβουμε την ίδια μεθοδολογία το ανοιχτό ή το σύστημα επιπαντός επιστητού. Λέω να εστιαστούμε σε δύο-τρεις προκλήσεις και αυτές να αντιμετωπίσουμε. Όχι όλα ανοιχτά. Και γιατί να μην ανατρέξουμε ακόμη και στον ύμνο μας, ακόμη και στη σημαία. Δεν νομίζω όμω ότι είναι παραγωγικό κάτι τέτοιο να επαναλάβουμε πράγματα που ήδη έχουμε πει στο παρελθόν. Καλύτερα να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Έτσι θα έχουμε και την ευκαιρία να προωθήσουμε τις προτάσεις μας και να ευοδοθούν αυτές οι απόπειρες. Πιστεύω ότι όπως είπαν και, ο κύριος Μπρό και η κυρία Μπρέσο, ε, είπαμε ότι δεν έχουμε οικονομική διακυβέρνηση γενικώ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Γιατί η συνέλευση δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα αυτό. Όλοι παρέμεναν στη συνθήκη του Μάστριχτ που έλεγαν αυτή είναι η συνθήκη του Μάστριχτ, ας μην προσθέσουμε τίποτα. Εν τω μεταξύ όμως ανέσκυψε ε, η χρηματοπιστωτική κρίση, η οικονομική κρίση και άλλαξε η καθημερινότητά μας και διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν αρκετά όλα αυτά που είχαμε και δεν νοείται η Οικονομική και Νομισματική Ένωση χωρίς Οικονομική Ένωση, Φορολογική, Δημοσιονομική Ένωση, Κοινωνική Ένωση. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια απάντηση για όλα αυτά τα ερωτήματα. Και σίγουρα κάποια θέματα μπορούμε να τα λύσουμε εντός της συνθήκης. Όχι όμως και τα πάντα. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Επίσης, μπορούμε να ενσωματώσουμε διάφορες πολιτικές και μηχανισμούς που θεσμοθετήθηκαν εκτός της συνθήκης. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ο μηχανισμός σταθεροποίησης. Γιατί αυτά ξεπερνούν και το σύμφωνο σταθερότητας και τη συνέλευση. Ήταν πράγματα που αναδύθηκαν εξαιτία της κρίσης και με διακυβερνητικούς μηχανισμούς. Θα πρέπει όλα αυτά να τα επαναφέρουμε στο σύστημα. Και επίσης να ορίσουμε τι εστί οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκρισταλώσει τη θέση του γι' αυτό και έχει υπερψηφίσει πολλά ψηφίσματα που διατρανώνουν τη δική μας θέση για το τι εστί οικονομική διακυβέρνηση. Βέβαια, προς το παρόν το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι τέσσερις πρόεδροι, γιατί το πρώτο έγγραφο ε, που είδαμε από τον Ζαν Κλον Γιουνκέρ θέτει 11 ερωτήματα. 11 θεμελιώδη ερωτήματα για τα οποία ε, είχαμε δηλώσει ανέκαθεν στο Κοινοβούλιο ότι θέλουμε σύγκληση, θέλουμε να ξεπεράσουμε το συντονισμό των πολιτικών, θέλουμε να επεκτείνουμε τις ε, δημοσιονομικές πολιτικές Υπάρχουν όμως ακόμη κάποια εμπόδια, κάποια φραγμή λόγω της συνθήκης, ακόμη και στην εσωτερική αγορά και στις πολιτικές μας της εσωτερικής αγοράς. Για παράδειγμα, Ενεργειακή Ένωση. Όταν υποβάλλουμε τις ιδέες μας για την Ενεργειακή Ένωση, λέει ένας δημοσιογράφος, ε, ναι, το τάδε άρθρο της συνθήκης λέει ότι η ενεργειακή πολιτική αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Όντω. αλλά δεν μπορούμε ταυτόχρονα να θέλουμε να δημιουργήσουμε ενεργειακή ένωση και να ε, βαλτώνουμε σε τέτοιου είδη συζήτηση. Κεφαλαία αγορά, τελωνιακή ένωση, τραπεζική ένωση, εσωτερική αγορά. Θέλουμε να τις προωθήσουμε, αλλά ακόμα υπάρχουν ε, εμπόδια στην συνθήκη που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη και σχεδόν τις προτάσεις αυτές ανέφικτες. Οπότε πρόκειται για ένα ευρύτερο εγχείρημα που χρειαζόμαστε. Ένα εγχείρημα στο οποίο ε, σχεδόν και παρά τη θέλησή μας και λόγω της κρίσης. Οπότε τώρα πια ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση και να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του τι είναι εφικτό εντός της συνθήκης, στο πλαίσιο της συνθήκης και τι θα πρέπει να γίνει εκτός της συνθήκης. Δεύτερη πρόκληση θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ε, εγκαθίδρυση ενός ε, γνήσιου δημοκρατικού συστήματος και λογοδοσίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί εκεί έχουμε ακόμη ελλείμματα. Συνεχίζω αυτό που είπε ο Έλμαρ Μπρόκ. Το ισχύον σύστημα όχι μόνο είναι περίπλοκο, αλλά δεν είναι και πολύ ορθολογικό. Βέβαια αυτό δεν μας εμποδίσει ε, στην πολιτική, το, η έλλειψη ορθολογισμού, αλλά μερικές φορές μπορεί να μας δημιουργεί δυσκολίες. Γιατί δεν έχουμε ε, ένα πλήρες ε, εκτελεστικό σώμα με δύο νομοθετικές εξουσίες που το ελέγχουν. Ίσως θα μπορούσαμε αυτή την πορεία να ακολουθήσουμε. Προς το... Έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προς το παρόν είναι θεσμικό όργανο. Δεν ξέρω αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση. Εν πάση περιπτώσει άλλο θέμα αυτό. Αλλά υπάρχουν ακόμη αδυναμίες. Γιατί ε, το Συμβούλιο έχει ταυτόχρονα και νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες. Πού, βλέπω, πού συναντούμε κάτι τέτοιο, σε ποια νομή τάξη, πουθενά συσσόρευση στον ίδιο φορέα εκτελεστικών και νομοθετικών εξουσιών. Κάτι τέτοιο δεν ευδοκιμεί σε ένα κανονικό νομικό σύστημα. Και ο τρόπος της Προεδρίας είναι παράλογος. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με μόνιμο πρόεδρο. Έχουμε τα Συμβούλια. Έχουμε την Εκπεριτροπής Προεδρία. Έχουμε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι παρόν. Έχουμε το Eurogroup, ε, μια ομάδα εντός της, ε, του, του κανονικού συμβουλίου, με επίσης πρόεδρο. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Λύσεις δεν έχουμε, αλλά τουλάχιστον τις ερωτήσεις να τις θέσουμε. Θα συνεχίσουμε με αυτό το πλαίσιο ή μήπως όπως είπε ο Έλμαρ στην εισαγωγή του ήρθε η ώρα να έχουμε ένα πιο φυσιολογικό σύστημα μιας εκτελεστικής εξουσίας και δύο σκελών της νομοθετικής εξουσίας που θα ελέγχουν την μία ενιαία εκτελεστική εξουσία. Και ο ένας βραχίωνας της νομοθετικής εξουσίας να εκπροσωπεί τους λαούς και ο άλλος τα κράτη. Επίσης, άλλες προκλήσεις. Είμαι στην ομάδα υψηλού επίπεδου για, τη, για τους ίδιους πόρους. Το θέμα της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης σημαντικό. Βέβαια, εδώ υπάρχει μεγάλη προεργασία και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την ομάδα υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους. Αυτά όμως θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη γιατί χρειάζονται σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Είμαστε το μόνο κοινοβούλιο που αποφασίζει μόνο για τις δαπάνες και όχι για τα έσοδα. Συνήθως τα κοινοβούλια το αντίθετο έργο έχουν. Αποφασίζουν για τα έσοδα και για τις δαπάνες. Εμείς είμαστε η μόνη βουλή που έχουμε το ίμιση των αρμοδιοτήτων ενός κανονικού κοινοβουλίου. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, αλλά θα το αναφέρω. Το Spitzenkandidaten, αυτές οι προτάσεις για έναν επικεφαλής ε, για την Προεδρία της Επιτροπής των Κομμάτων. Θα συνεχίσουμε αυτή τη μέθοδο, θα την ευαθύνουμε ή όχι. Μήπως χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό ε, ψηφοδέλτιο με τέτοιους Spitzenkandidaten. Ιδέες πολλές, αλλά ούτε μία έκθεση στην Ολομέλεια σχετικά. Και επίσης, το μέγεθος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μήπως και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Γιατί χρειαζόμαστε μια νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το θέμα αυτό πριν το 2019. Πριν την επόμενη σύσταση δηλαδή της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και άλλες πολιτικές, θεμελιώδεις αξίες. Γνωρίζουμε ότι οι διατάξει της ηθίκη δεν είναι και πολύ αποτελεσματικέ για το θέμα αυτό. Μήπως θα πρέπει να τις αναθεωρήσουμε και με ποιο τρόπο. Και τέλος, ε, η διάσκεψη των Προέδρων και ο πρόεδρο ε, μα ζήτησε στο θέμα αυτό να ασχοληθούμε και με το θέμα της ενιαίας έδρας, αντί να συντάξουμε ξεχωριστή έκθεση για την ενιαία έδρα. Να το αναφέρουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί θέλουμε να επιλύσουμε το θέμα της ενιαίας έδρας και εδώ χρειαζόμαστε προηγούμενη αναθεώρηση της συνθήκης. Τρίτον, τρίτη πρόκληση που είναι συνειφασμένη με το βρετανικό ζήτημα. Πού μπορούμε να φτάσουμε, δηλαδή να, εξαιρείται, να αυτοεξαιρείται ένα ε, ένα κράτος από διάφορες πολιτικές και ταυτόχρονα είναι πλήρες μέλος της Ένωσης και όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Αν κανείς επιλέξει ρήτρα αυτοεξαίρεσης ε, για διάφορες πολιτικές, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Ποια είναι τα όρια αυτής της αυτοεξαίρεσης. Μερικοί λένε θέλουμε δύο είδη με κρατών μελών, δύο κατηγορίες κρατών μελών. Ίσως και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε στο μέλλον, στα πλαίσια της έκθεσης. Μήπως ε, ευκαιρία θα πρέπει να λύσουμε και το θέμα της λογοδοσίας των πολιτικών της Ευρωζώνης. Μήπως θα πρέπει επευκαιρία της έκθεσης αυτής να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της πληθώρας των ενώσεων που έχουμε εντός της Ένωσης, γιατί έχουμε την, την ε, Ένωση του Ευρώ, του Σέγγεν, των εσωτερικών υποθέσεων, του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Για κάθε πολιτική έχουμε και διαφορετική ένωση. Πολύ περίεργο όν αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολιτικές που τα κανονικά μέλη ε, δεν, της Ένωσης δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν, ενώ, μέλη, ενώ χώρες εκτός της Ένωσης υποχρεούνται να συμμετέχουν. Πώς είναι δυνατόν να απαλλάσσουμε χώρες από συμμετοχή στο Σέγγεν και να ε, εντάσσουμε στο Σέγγεν χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, έχουμε εδώ ένα πολλαπλασιασμό των ενώσεων με τέτοιου είδους πολιτικές, γιατί κάθε ρήτρα αυτοεξαίρεσης και κάθε ρήτρα προαιρετικής ένταξης και κάθε εξαίρεση είναι μία νέα παρέκκληση από το φυσιολογικό σύστημα μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα ενιαίο πλέγμα πολιτικών. Και τέλος, για το βρετανικό ζήτημα και αυτό το θεσμικό πλαίσιο, δεν ξέρω αν είναι η ώρα να προβλέψουμε και μια γενική πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και όχι μόνο για τα ζητήματα που σήμερα προβλέπονται, αλλά και για οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, για θέματα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Το συζητήσαμε ήδη στην Επιτροπή μας σε προηγούμενες εκθέσεις. Και τέλος, η γεωπολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλη πρόκληση. Βλέπετε τι συμβαίνει στα σύνορά μας στην άμεση γειτονία μας. Μήπως τώρα θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε ένα ποιοτικό άλμα και ως προς τη γεωπολιτική μας σημασία. Νο, νόμιζα ότι το 94 ήταν η χειρότερη χρονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ βέβαια γεννήθηκα το 93, αλλά δεν είμαι εγώ ο Το 94 όμως, όταν η, Εθνική, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση αποφάσισε να πει όχι σε ένα σχέδιο που είχε σχέση με την ε, άμυνα, την ε, Ένωση για την Άμυνα αλλά και την Πολιτική Ένωση γιατί χρειαζόταν Πολιτική Ένωση για να πραγματοθεί η Αμυντική Ένωση. Νομίζω ότι ήταν ε, αποφράδα χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994. Επίσης, ε, εξακολουθεί να ισχύει ομοφωνία για τα περισσότερα θέματα πολιτικής. Ακόμη, χθες ο πρόεδρος Τάσκ αυτό είπε στην Ολομέλη. Ότι θα ήθελε να προωθηθούν κάποιες πιο δραστήριες πολιτικές στις εξωτερικές υποθέσεις, αλλά κάτι τέτοιο είναι αδύνατο γιατί θα πρέπει οι αποφάσεις να ληφθούν με ομοφωνία. Ίσως κάποιες ρήτες πασαρέλας ε, στην εξωτερική πολιτική. Γιατί όχι. Και το θέμα της ε, κοινότητας της άμυνας ή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Άμυνας και πώς θα την προωθήσουμε για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο απορίες έδωσα, μόνο ερωτηματικά έβαλα. Και τώρα πώς θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Ε, και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Με συνέλευση, ναι ή ου. Και με ποιο άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει το σημερινό μου μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να εστιαστούμε σε αυτές τις τέσσερις ειδικέ προκλήσεις τέσσερα συγκεκριμένα ζητήματα. Και να μην ε, ξαναρχίσουμε μία ανοιχτή συζήτηση επί παντός επιστητού, όπως είχε γίνει μερικές φορές στο παρελθόν. Ευχαριστούμε θερμός, Γκί. Έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο να με ενημερώσετε, γιατί έχω ήδη σημειώσει κάποιους. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη που... Ραμόν Χαουρέγγι. Θα ήθελα καταρχάς, ε, Πρόεδρε, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συζήτηση που ξεκινήσαμε. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ύπαρξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση αυτή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε αυτά που πρέπει να δούμε και πιστεύω απόλυτα ότι μια συνθήκη που έχει μόνο πέντε χρόνια ζωής αντιμετώπισε παρόλα αυτά τρεις εξαιρετικές περιστάσεις κρίσιμες που απαιτούν τώρα αποφασιστικές κινήσεις. Έχουμε μια τεράστια χρηματοπιστωτική κρίση, έχουμε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση στο γεωπολιτικό πλαίσιο έχουμε μια άμεση ανάγκη προσαρμογής της δημοκρατίας μας σε μια Ευρώπη που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνα ευρωσκεπτικιστή. Κι, με συγχωρείτε. Και θυμίζω ότι αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που έχουμε. Δηλαδή ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο, πλάνο, όπως αυτό που σκιαγράφησαν οι προαλήσαντες που είναι λαμπροί συνάδελφοι και που είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουν σε ένα πρώτο σχέδιο κειμένου εξαιρετικό πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα πλαίσιο πολιτικό που δεν είναι καθόλου γόνιμο για τέτοιου είδους φιλόδοξες αλλαγές. Δεν μπορώ να φανταστώ ρεαλιστικά πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν τόσο φιλόδοξες αλλαγές σε αυτό το πλαίσιο το τωρινό, το υφιστάμενο, αυτό που ζούμε. Θυμάμαι στο τελευταίο συμβούλιο που ο κύριος ε, Σούλτς ο ίδιος μιλώντας σχεδόν εκ μέρους του, συνόλου του Ευρωκοινοβουλίου έλεγε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αναθεώρηση συνθήκης, συνθήκων. Δηλαδή, το βασικό ερώτημα είναι τι κάνει το Ευρωκοινοβούλιο σε μια τέτοια χρονική στιγμή. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν σωρία από πράγματα που δεν λειτουργούν καλά. Επομένως, ε, καταρχάς χρειαζόμαστε μια διάγνωση όλων εκείνων που βλέπουμε, και είναι πολλά, που δεν λειτουργούν καλά, τα ανέφεραν και οι συνάδελφοι, θα πρέπει σαφέστατα να πούμε στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, στα κόμματα, στα εθνικά κοινοβούλια, τι εμείς βλέπουμε που να πάσχει για να έχουμε ή δυνατόν μια κοινή διάγνωση και από εκεί και πέρα τι θα μπορούσαμε κοινώς να προβλέψουμε ώστε να επαναρθώσουμε την κατάσταση αυτήν. Και μπορούμε να σκεπτόμαστε μια δυνητική τροποποίηση των συνθήκων αλλά ας τοποθετήσουμε ένα πλαίσιο, ας δώσουμε κάποιες ενδείξεις. Αντί να επικαλούμαστε ε, εξαιρετικά φιλόδοξα πράγματα. Ας, προσπαθήσουμε να εστιαστούμε σε πράγματα στα, τα οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε σε αυτήν εδώ την εντολή και όχι στο μέλλον. Ευχαριστώ, Ιωλάινεν. Εγώ θεωρώ για τις δύο αυτές εκθέσεις πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη για τη λειτουργικότητα και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οπωσδήποτε αν δει κανείς την κατάσταση και η Κομισιόν ε, και το Συμβούλιο έχουν παραλύσει και μόνο εμείς ε, θα κάνουμε αυτή την συζήτηση για το όραμα και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μεταφέρουμε αυτή τη συζήτηση προς τα έξω. Το πρωί συζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που συζητάνε αυτά τα πράγματα και θα επιτύχει αυτό το θέμα μόνο εάν τους συμπεριλάβουμε και αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν να εξαντλήσουμε το δυναμικό της συνθήκης Λισαβόνας. Θα αναφέρω μόνο τη χρηματοδότηση της Ένωσης που είναι ελληματική, τι θα γίνει με τους ίδιους πόρους, τη δημοκρατική αρχιτεκτονική της Ένωσης και βεβαίως ε, τα ελλείμματα που έχει η συνθήκη του Μάστριχτη. Πραγματικότητα πλέον δεν ανταποκρίνεται αυτό, σε αυτό το οποίο είχαν φανταστεί πριν από 25 χρόνια στο Φάστριχτ. Βλέπω πως ο Γκίφερ Χόφστατ περιορίζεται σε τέσσερα θέματα Οπότε το ερώτημα είναι αν θα περιοριστούμε ή αν η επόμενη συνέλευση θα προσπαθήσει να κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κόσμος έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Α, οι σοσιαλιστές Μιλάνε μάλιστα. Λοιπόν, ξεκίνησα. Νομίζω πως ε, οι συνθήκες ε, έχουν ε, αποδειχθεί πολύ πιο ευέλικτες από ό,τι περίμενε πολλοί κόσμος. Προχωρήσαμε πολύ στην Νομισματική Ένωση και σε άλλα ζητήματα με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες και δεν έχουμε ακόμα εκμεταλλευτεί πλήρως ε, πράγματα όπως η ενισχυμένη συνεργασία, η μόνιμη δομημένη συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής κτλ. Ο Έλμαρ ανέφερε πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν με αλλαγή της συνθήκης αλλά μπορούν και χωρίς η εσωτερική οργάνωση του Συμβουλίου, ένας επίτροπος ε, να προεδρεύει στο Eurogroup η μεταρρύθμιση της διαδικασίας του τριμερούς διαλόγου. Αυτά δεν χρειάζονται αλλαγή της ε, συνθήκης. Όταν ε, μιλάμε για τη σημαία και τον ύμνο, είναι αδιάφορο αν θα είναι στην συνθήκη ή όχι. Επίσης ε, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό να πάει κανείς να δει το Ryder Cup, το Ryder Cup στο Golf και βλέπουν, ε, βλέπουμε διάφορους ευρωσκεπτικιστές με το ευρωπαϊκό σημαίακι βεβαίως γιατί οι ομάδες είναι Ευρώπη και Αμερική. Έτσι προωθείται η χρήση της σημαίας και όχι με το να το γράψουμε στη συνθήκη. Ε, τώρα, ότι μπορούμε να αλλάξουμε χωρίς την αλλαγή της συνθήκης, σε πολλές περιπτώσεις ούτως ή άλλως δεν υπάρχει η απαραίτητη συνένεση είτε μιλάμε για ευρωομόλογα πλήρως ανεπτυγμένα με κοινό εθνικό χρέος ή να περάσουμε στην ε, ειδική πλειοψηφία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να φανταστούμε που μπορεί να τα θέλουμε ή όχι, αλλά δεν υπάρχει συνένεση ούτως ή άλλως. Παραμένει το θέμα των ε, διακυβερνητικών συνθήκων. Την... Η συνθήκη ας πούμε για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο έγινε διακυβερνητική ε, όχι επειδή το θέλαμε αλλά γιατί κάποιο κράτος ε, το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή προέβαλε βέτο. Αυτό το οποίο έκαναν όμως ανταυτού ήταν να δημιουργήσουμε μία ξεχωριστή συνθήκη η οποία ε, πήγαινε όσο δυνατόν πιο κοντά στις υφιστάμενες. Πράγματι, Γκί, δεν είναι λογικό αυτό το σύστημα. Η χώρα μου έχει και ένα εθνικό πολιτικό σύστημα που δεν είναι πάρα πολύ λογικό με μια βουλή των Λόρδων, με εκχώρηση ε, τοπικών εξουσιών στην ε, Βόρεια Ιρλανδία, Σκοτία, Ουαλία, αλλά όχι στην Αγγλία, δεν είναι πολύ λογικό. Αλλά μπορεί να διατηρηθεί, ειδικά εάν ο κίνδυνος της αλλαγής είναι μεγαλύτερος από τους ε, κινδύνους της διατήρησής του. Ναι, είναι χώρες που έχουν μείνει πίσω, παραδείγματος χάρη Κύπρος, Ιρλανδία, Βρετανία δεν είναι στο Σέγγεν, άλλες χώρες δεν είναι στο ευρώ. Άλλε δεν είναι στο δικαστήριο για τα διπλώματα βρεστιχνίες. Πάντα είναι μια μειοψηφία, καμιά φορά και μια χώρα μόνη της. Είναι διαφορετικοί οι συνδυασμοί αναλόγως στο θέμα. Τώρα αν είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά μοιραίο για την Ένωση, όχι εγώ θεωρώ πως ε, απλά είναι κάτι που πρέπει να δεχτούμε αυτή τη στιγμή και θα ξεπεραστεί έναν καιρό. Δεν είναι ζωτικό. Τέλος, οι αναφορέ για, το βρετανικό ζήτημα. Ας περιμένουμε τι εκλογέ το Μάιο να δούμε πώ έχει το βρετανικό ζήτημα, αν υπάρχει βρετανικό ζήτημα. Πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των εκλογών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, πρέπει να συντομεύουμε γιατί ε, περιμένουμε. Ευχαριστώ. Είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της συνθήκης και μπορώ να πω ότι είμαι κάπως απογοητευμένος γιατί νομίζω ότι θα σημειώναμε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο αν είχαμε ήδη συγκεκριμένες προτάσεις ε, των εισηγητών. Γιατί είναι κάπως χαοτική μεθοδολογία που υιοθέτησαν. Ο κύριος Φερχόφσταν είπε ότι η θεσμική γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπλοκη. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Και το πρόβλημα έγκυται στο να ε, υποβάλουμε συγκεκριμένες χειροπιαστές ε, θετικές προτάσεις που θα βελτιώνουν και θα πλουστεύουν αυτή την γεωγραφική περιπλοκότητα. Και από τη στιγμή που οι εισηγητές δεν υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις, τότε θα είμαστε συνέχεια στο σημείο 0. Ε, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ. Γι' αυτό και θα ήθελα να το ρωτήσω γιατί είπατε ότι υπάρχει δυνατότητα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει και πρόεδρος του Συμβουλίου. Έτσι κατάλαβα τουλάχιστον. Μπορείτε να αναπτύξετε κάπως αυτή σας τη σκέψη. Γενικώ πάντως, θα σας παρότρινα να περάσουμε από την γενική και όριστη συζήτηση στη συγκεκριμένη συζήτηση επί αυτών προτάσεων. Νομίζω ότι έτσι θα διευκολύνει καλύτερα και το έργο μας μια τέτοια συγκεκριμένη υποβολή προτάσεων. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί καταφθάνουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Σίγουρα θα συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι περιμένουν ε, τα έγγραφα με συγκεκριμένες προτάσεις. Καλό θα ήταν όμως και πριν ε, την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων να γίνουν κάποιες συζητήσεις πρώτα. Πάντως ε, θα έχουμε, θα έχουμε και έγγραφα. Σας ευχαριστώ. Θα, θα περιοδικά σε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά πριν απαντήσω στην ερώτηση. Εντάξει. Ich möchte die Frage, gestellt να πω δύο λόγια για τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι και για το ανακοινωθέν του τύπου στην Πολωνία. Εγώ φαντάζομαι πως καλός πρόεδρος θα ήταν ο Ντόναλτ Τούσκ, αλλά και ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ. Οποιοςδήποτε από τους δύο δηλαδή. Αυτό για να μην φέρω σε αμηχανία τον κύριο Τούσκ. Σας ευχαριστώ. Εντάξει συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους ε, τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ε, συζήτηση αυτή. Έχουμε τώρα τη συνάντηση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρακαλώ να καθίσετε.